Καλό σα απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε. Good afternoon, dear colleagues. Καλό σα απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Please be welcome. ορίσατε λοιπόν στη συνεδρίαση αυτή τη Επίτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και πάλι. Και με ένα βαρύ φορτίο εργασία στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο λοιπόν σημείο. Είναι η έγκριση τη ίδια τη ημερήσια διάταξη φυσικά. Κάποιες αλλαγές έχουν εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη. Σημειώστε ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τα σημεία 6 έως 11 έχουν αλλάξει οι προθεσμίες αυτές από 29 Σεπτεμβρίου 18.00 το σημείο 30 στις 29 Σεπτεμβρίου 18.00 το σημείο 30 αναβάλλεται στην επόμενη συνεδρίαση το 31 επιβεβαιώνεται το σημείο 32 αναβάλλεται και αυτό το σημείο 2 αναγγελίες προαναγγελίες Προέδρου ανακοινώσεις δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση για τα προηγούμενα συμφωνείτε με τα όσα σας πρότεινα με το σημείο 1, έγκριση ημερήσια διάταξη. Εγκρίθηκε λοιπόν η ημερήσια διάταξη έτσι. Σημείο 2, ανακοινώσει Προέδρου. Απλά να σα υπενθυμίσω εδώ κάτι, ότι το ψήφισμα της Ευρωβουλής ε, <clears throat> για το μέλλον πρόγραμμα τη Στοκχόλμη, ήδη τον Ιούλιο αποφασίσαμε να εγγράψουμε μια κοινή πρόταση ψηφίσματος με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και Νομικών Θεμάτων και την άλλη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σε σχέση με το άρθρο 51 των κανονισμών του Κοινοβουλίου. Θα έχουμε κοινέ συνεδριάσει σχετικά στη συνέχεια και ζητώ από όλου σας να επικαιροποιήσετε την ημερήσια διάταξη έτσι. 8 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες παρουσίαση του σχεδίου ψηφίσματος. 12 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα. Το δικό μας ψήφισμα θα υποβληθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια κατά την κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση που σχεδιάζεται για την 16η-17η Νοεμβρίου. Ψήφιση θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια του, της Ολομέλειας η περίοδου συνόδου του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Θα βρείτε το χρονοδιάγραμμα, έχει διανεμηθεί. Και σε σχέση λοιπόν με ε, την έγκριση του χρονοδιαγράμματος για το 2010 που υιοθετήθηκε στην τελευταία συνεδρίασή μας, δεν υπάρχουν σχόλια σχετικά, δεν υπάρχουν. Περνάμε στο 3, σημείο 3 που είναι οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου σε σχέση με τις συστάσεις για συντονιστές και ορισμό εισηγητών. Ε, προτάσεις, ε, συστάσεις συντονιστών για τον ορισμό εισηγητών. Οι συντονιστές συνήθαν, συναντήθηκαν για αυτό το σκοπό και έχουμε τις εξής, ε, τους εξής διορισμούς ως εισηγητών. Πρόληψη και καταπολέμηση ανθρώπινου εμπορίου και προστασία θεμάτων. Η η κυρία Άννα Χέγγ. Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία. Η η συγγήτρια η κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη. Η υπηρεσία για την διαχείριση και διαχειριστική αντιμετώπιση μεγάλων συστημάτων IT μεγάλης κλίμακας για την διαχείριση SIS Schengen Information Service 2 και VIS Visa Information System εισηγητής ο κύριος Καύλος Κουέλιο δημιουργία διαμεσολαβητών και υπηρεσιών γραφείων διαμεσολαβητών σε σχέση με liaison officer, εισηγητής διεθνεμέρα. Σε σχέση με ποινικέ διαδικασίες, ποινική δικονομία, εισηγήτρια κυρία Σάρα Λάρφορντ. Πειραματικά εργαστήρια ιατροδικαστικής, ο κύριος Τίμωθη Κέρκοπ η εφαρμογή κανόνων όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τέρου συμπεριλαμβανομένης και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίε και δεδομένα η συγγήτρια η κυρία Σόφι Ιντφέλτ πίνακα, κατάλογο τρίτων χωρών που οι πίκοοι του υποβάλλονται σε εξαίρεση από θεωρησει διαβατηρίων στο πέρασμα συνόρων η κυρία Τάνια η συγγήτρια δημιουργία μιας, ενός δικτύου πρόληψης εγκλήματος πανευρωπαϊκού, η συγγήτρια Σόνια Αλφάνο. Περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Ζιμπάμπουε. Η συγγητής ο κύριος Λουί Μισελ. Δεν υπάρχουν σχόλια για τους διορισμούς, ενστάσεις, αντιρρήσεις. Εσείς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών 20 περίπου προτάσεις είχαμε για γνωμοδοτήσεις ή εκθέσεις. Ναι, Πρόεδρε, έλεγα ότι στην τελευταία συνάντηση συντονιστών είχαμε 20 περίπου πάνω κάτω θέματα που είχαν προταθεί για γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις. Καταλήξαμε σε 10 περίπου. Ήδη έχουν διοριστεί οι συγητές σχετικά. Όμως έθεσα τότε στο παρελθόν ένα ερώτημα και αυτό εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων μελών στην Ευρωβουλή ώστε να έχουμε δύο συγκεκριμένες ε, εκθέσεις ε, δραστηριότητες ε, της Frontex για το, την Ελβετία και το Liechtenstein και σε σχέση με μέτρα εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων όσον αφορά την κατάσταση στη Σομαλία θα ήθελα να πω ότι δεν άκουσα τίποτα παραπέρα για αυτά τα θέματα. Αν όμως είμαι σωστά πληροφορημένος, στη συνάντηση των συντονιστών είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία. Δηλαδή, εκθέσεις που δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον κάποια ομάδα για αυτές θα επιστρέφουν σε ένα κοινό συλλογικό ας το πούμε έτσι pool και θα μπορούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι να τις ζητήσουν θα ζητούσαμε εξ ονόματο και μας ενδιαφέρει εξ ονόματο των μη εγγεγραμμένων να πάρουμε αυτέ τις δύο εκθέσει. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει πρακτικά με αυτέ τι δύο προτάσεις για εκθέσει. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, λέει ο Πρόεδρος, να σας ενημερώσω ότι αύριο αυτό το σημείο θα συζητηθεί ακριβώς στη συνάντηση των συντονιστών στις 9 το πρωί, 9.00. Τι θα κάνουμε με τις εκθέσεις και τα μόρια, τους πόντους, όταν θα έρχεται η ώρα των κοινοβουλευτικών ομάδων ή και των μη εγγεγραμμένων να επιλέξουν. Αυτό το σημείο θα συζητηθεί λοιπόν αύριο στις 9 το πρωί, εντάξει. Και θα προσκληθείτε κι εσείς να συμμετάσχετε και θα εισακουστείτε. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες, ε, άλλα σχόλια, παρατηρήσεις, θα συνεχίσουμε λοιπόν στο σημείο με το σημείο 4. Δημιουργία μιας υπηρεσίας υποστήριξης για θέματα ασύλου στην Ευρώπη. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Και το τι γίνεται σχετικά. Θα ξεκινήσουμε σήμερα για την ίδρυση της υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο που είναι σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Ο κ. Ζων Λαμπέρ είναι από πλευρά μα εισηγητή. Γι' αυτό το, ε, την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στις 7 Μαΐου είχαμε εγκρίνει μια πρόταση ε, για έγκριση από την Ευρωβουλή με τροπολογίες. Είναι συναπόφαση αυτό το δελτίο. Βρισκόμαστε σε δεύτερη ανάγνωση τώρα. Το χαρτοφυλάκιο είναι, έχει προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία όπως όλοι θα γνωρίζετε. Τυπικές και επίσημες επαφές υπάρχουν μεταξύ εισηγητού Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις που δημιουργούν μια υπηρεσία που θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη σε σχέση με θέματα που αφορούν την το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου. Είναι ένα από τα κυριότερα θέματα που αναφέρεται στο πρόγραμμα σχετικά. Και ενδιαφέρεται να υπάρξει συνεργασία εισηγητής με μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και τους σκιώδης εισηγητές ιδιαίτερα. Του του τώρα αυτό που θα κάνω είναι θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή που καλείται τώρα να παρέμβει. Ναι, να κάνει η κυρία Λάμπερ την παρουσίασή τη, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω προαναφέρθηκε πριν, αυτό είναι μια έκθεση όπου το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Τώρα βρισκόμαστε στην διαδικασία ω Ευρωβουλή τη συζήτηση, των συζητήσεων με τη Σουηδική τώρα Προεδρία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οπωσδήποτε φυσικά και με του σκιώδει εισηγητέ, που του ευχαριστώ πολύ για την, το, την εργασία τους και το ζωντανό ενδιαφέρον τους για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ως ένα πακέτο, μια δέσμη αντιμετωπίζουμε τα μέτρα τα οποία αφορούν το Δουβλίνο, τη Eurodac, τους όρου υποδοχής και αποτελεί αντικείμενο σκέψεων αυτή τη στιγμή. Αν θα συνεχίσουμε με το πακέτο αυτό ή αν θα βρούμε σημαντική συμφωνία με το Συμβούλιο και προχωρήσουμε ταχύτατα επ' αυτού. Κατανοούμε το ενδιαφέρον του Συμβουλίου για τα κράτη και των κρατών μελών να σημειωθεί πρόοδος σίγουρα, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει η σωστή διαδικασία και ότι θα διασφαλιστούν τα θέματα της υπηρεσίας ε, υποστήριξης για το άσυλο με τον σωστό τρόπο ο ρόλο αυτού του γραφείου υποστήριξη είναι να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή, στην εκτέλεση του κεκτημένου για τα θέματα ασύλου που ήδη υφίσταται και να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση που θα επιτευχθεί. Η Ευρωβουλή θέλει να υπάρξει βελτιωμένη ποιότητα, αναβαθμισμένη ποιότητα όσον αφορά την λειτουργία του συστήματο για χορήγηση ασύλου ω έχει σήμερα με βελτιώσει στο μέλλον. Τρίτο τμήμα να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σημαντική ξεχωριστή πίεση λόγω γεωγραφικής τους ίσως θέσης ή λόγω άλλων συγκεκριμένων ιδιομορφιών. Θέλουμε πάρα πολύ να, με σθένος να διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη. Να θυμόμαστε όμως από την άλλη πλευρά ότι είναι και μέρος και τμήμα των ιδίων των ευρωπαϊκών διαδικασιών και διεργασιών. Και δεν είναι απλά ένα διακυβερνητικό σώμα, αλλά τμήμα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα θέματα για μας που τώρα εντοπίζονται και ταυτοποιούνται στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο προέρχονται φυσικά και λογικά από τροπολογίε που εγκρίθηκαν σε σχέση με την Ευρωβουλή, όπω προαναφέρθηκε το Μάιο 2009 εφέτο. Μια-δυο αφορούν τη δομή, τη διάρθρωση του ε, Γραφείου τη Υπηρεσία ε, Υποστήριξη για το Άσυλο και κυρίω ποιο θα είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό το γραφείο. Αυτό που ζήτησε η Ευρωβουλή είναι να έχουμε σημαντικό λέγην στην απόφαση να συνεπηρεάζουμε για την επιλογή του Προέδρου του διοικητή και σε σχέση με το shortlist για την παρουσίαση σε σχέση με το κοινοβούλιο φαίνεται ότι όμως το Συμβούλιο έχει δυσκολίες να δεχθεί αυτό το αίτημα. Ζητούμε επίσης να μπορεί να ζητήσει την σύνταξη εκθέσεων από την Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου το Κοινοβούλιο για θέματα του κεκτημένου και για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης επίσης όσον αφορά την έκθεση που θα συντάσσεται από την υπηρεσία αυτή προ την Ευρωβουλή. Φαίνεται ότι και αυτά τα αιτήματα δημιουργούν κάποιες τριβέ ή δυσκολίε για κάποιου περίεργους λόγους στο Συμβούλιο. Σημαντικό είναι επίση για μας να δούμε τον ρόλο του διαβουλευτικού συμβουλευτικού φόρουμ που μη κυβερνητικέ οργανώσει, μη κοιό, ε, συναθρίζει που ε, λειτουργούν μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Συμφωνήσαμε, είχαμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο ότι θα βλέπαμε την ιδέα για την κοινωνία των πολιτών, civil society, γιατί είναι σημαντικό οι τοπικές αρχές να δρουν σωστά, όχι μόνο για τους όρους υποδοχής των ασυλούχων, των ετούντων άσυλο, αλλά να μπορούν να εκφράζουν και τη φωνή τους μέσα σε αυτό το συμβουλευτικό φόρουμ. Κάποιο δρόμο πρέπει, πορεία να καλύψουμε ακόμα. Έχουμε αρκετό δρόμο να καλύψουμε για το πώς αυτό το ε, συμβουλευτικό φόρουμ θα δρά και τι θα κάνει διότι το αίτημά μας δύο φορές ετήσια να συνέρχεται δεν έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο ακόμα. Παρ' όλα αυτά έχουν διατηρήσει τον χαρακτήρα του διαβουλευτικού συμβουλευτικού αυτού φόρουμ αλλά όχι με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε εμεί. Είναι σημαντικό επίση για μα, ενώ είπατε η αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών θα εμπλέκεται για αυτά τα θέματα και αυτό δεν είναι τίποτα που εκπλήσει κανέναν. Αυτό είναι ο διεθνή θεσμό που είναι ο θέματοφύλακα αυτών των θεμάτων. Η διεθνή όμω ε, ε, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ε, είπατε αρμοστία για θέματα ασύλου πρέπει να επανεξεταστεί για να εγκριθεί. Και τώρα και το θέμα του, της δημιουργίας αυτού του γραφείου σε σχέση με τρίτες χώρες και για το ακριβώς πώς θα μπορεί να λειτουργεί και με ποια θέματα και σε ποια βάση. Νομίζω ακόμα θα έπρεπε διερευνητικά να δούμε τι επιθυμεί δέχεται το Συμβούλιο, ποιοι θα είναι οι όροι και οι διαχωριστικές γραμμές για αυτή τη συνεργασία ώστε να μην δώσουμε outsourcing, να μην γίνονται αλλού πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεισφέρουν στην αυθεντική λύση των προβλημάτων. Ένα τέταρτο θέμα είναι η υποστήριξη αυτή που θα πρέπει να δίνεται σε χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση, ιδιαίτερες πιέσεις ή τριβές και προβλήματα χώρες όπως η Μάλτα σίγουρα και ίσως μια-δύο χώρες ακόμα επιπλέον υπό του όρου των μηχανισμών αλληλεγγύη που λειτουργούν εκεί για αυτέ τι χώρε που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πίεση. Η Ευρωβουλή θεωρεί ότι κάτι σημαντικό και αποτελεσματικό πρέπει να γίνει. Υπάρχει υποχρέωση να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη με αλληλέγγυο τρόπο και όχι να λέμε δεκάρικου λόγου και να εκφωνούμε κάποιε εξαγγελίε για συνεργασία. Ακόμα διερευνούμε και αναζητούμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για αυτό το θέμα γιατί φαίνεται ότι κινείται το Συμβούλιο όλο και πιο μακριά προ μια βάση εθελοντική, εθελούσια συνεργασία Αυτά είναι τα θέματα. Δύο θέματα που αφορούν τη δομή, θέματα συμβουλευτικού φόρουμ, το εύρος και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ένα επιπλέον θέμα, και ένα θέμα έκφρασης αλληλεγγύης και μηχανισμού αλληλεγγύης. Ένας αριθμός άλλων θεμάτων όσον αφορά τις ομάδες υποστήριξης που θα έπρεπε να θελπιστούν και να λειτουργήσουν, πώς η πραγματογνωμοσύνη τους ε, θα προχωρεί. Εδώ είδαμε ότι και σε σχέση με την αποδοχή ε, τροπολογιών του Κοινοβουλίου σημειώθηκε πρόοδο. Καλοχαιρετίζουμε αυτή την πρόοδο από το Συμβούλιο. Υπάρχουν όμω θέματα που εκκρεμούν και αν θέλουμε γοργά να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό για αυτά τα θέματα, πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση, κίνηση από πλευρά του Συμβουλίου να ανταποκριθούν στα αιτήματά μα για να μπορέσει το τμήμα να, ε, για την υπηρεσία υποστήριξη ασύλου να τεθεί χωριστά από την γενική πολιτική για το άσυλο. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Λάμπερ. Κάποια μέλη ζήτησαν ήδη να παρέμβουν βέβαια. Πριν όμως γίνει αυτό, νομίζω καλό θα ήταν να ακούγαμε από την Προεδρία, τη Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου, από τον κύριο Λάρς Γιώχαν Λάνβακ, τα σχετικά. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Mr. Ο κύριος Λόμπακ λοιπόν έχει τον λόγο. Πρόεδρε σας ευχαριστώ θερμά. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε την ευκαιρία στην Σουηδική Προεδρία να σας προσφωνήσει ως μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και για αυτό το θέμα που πραγματικά είναι ένα θέμα που η Σουηδική Προεδρία δίνει σε αυτό ιδιαίτερη προτεραιότητα και σημασία. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη δύο φορές στο παρελθόν εκφράστηκε και τοποθετήθηκε για το κατεπήγον του να θεσπιστεί αυτό το γραφείο, αυτή η υπηρεσία πριν από τα τέλη αυτού του έτους, του ενεστώτος έτους 2009. Και ήταν σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα θέματα πρακτική συνεργασία, η υλοποίηση και εκτέλεση ενό κοινού ευρωπαϊκού συστήματο για τη χορήγηση ασύλου και η διευθέτηση θεμάτων ιδιαίτερη πίεση που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη θα πρέπει να είναι ακριβώ το έργο που θα επομιστεί αυτή η υπηρεσία. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες προηγούμενες ε, προημείο επαφές που έχουν γίνει ήδη. Και ήδη έχουμε πάρει μια εντολή, έχουμε λάβει εντολή μέσα στο πλαίσιο της Κορεπέρ. Είμαστε λοιπόν σε θέση με όλα αυτά να προχωρήσουμε σε άτυπους τριμερείς διαλόγους. Και μάλιστα με ένα πολύ σκόπιμο καρποφόρο αποτελεσματικό τρόπο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι με πολύ επικοδομητικό τρόπο αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτών των συζητήσεων στις οποίες προχωρούμε με την Ευρωβουλή παράλληλα με τις ε, γραμμές σίγουρα και συμφωνώ επ' αυτού για τα πιο σημαντικά, τόσο σημαντικά θέματα που η κυρία Τζιν Λάμπερτ προηγούμενα εξέθεσε. Απλά θα ήθελα να πω επ' αυτόν ότι ναι, μάλιστα, έχουμε πέρα από αυτά τα θέματα που λάβαμε υπόψη και αποδεχθήκαμε, έχουμε μια σειρά τροπολογιών επίσης που κατέθεσε η Ευρωβουλή όταν εκφράστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την πρόταση και τοποθετήθηκε σχετικά Σίγουρα λοιπόν θα εξετάσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα θέματα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από την Ευρωβουλή. Για παράδειγμα, τον διορισμό του εκτελεστικού διοικητή ή διευθυντή. Ήδη έχουμε αποδεχθεί κάποιες προτάσεις, κάποια στοιχεία από τις προτάσεις σας. Το βλέπετε, μπορείτε να το δείτε αυτό από το κείμενο της ίδιας της Κορεπέρ για την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, ε, UNHR κτλ. Και προσβλέπουμε σε μια σειρά ε, τέτοιων τριμερών ε, διαλόγων στο μέλλον τις επόμενες εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτού του χαρτοφυλακίου. Αποκινούμε την Ευρωβουλή. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστούμε κύριε Λόμπακ. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μουριέλ Γκίν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ μερικά για να τονίσω η σημασία προσδίδει ο Επίτροπός μας ο Ζακ Μπαγό σε αυτό το θέμα. Εμείς θα θέλαμε ομάδες εμπειρογνωμόνων να δημιουργηθούν στα κράτη-μέλη που θα υποβάλουν την αίτηση μέχρι το 2010. Θέλουμε η ανταλλαγή του, των καλών πρακτικών να γίνει το συντομότερο δυνατό μεταξύ κρατών μελών και κοινωνίας των πολιτών. Θα θέλαμε επίσης υπάρξει και η ανταλλαγή μεταξύ των διαφόρων αρχών που ασχολούνται με τα θέματα ασύλου. Στον επόμενο τρίλογο θα θέλαμε να διευκολυνθεί ένας τρίλογος μεταξύ των διαφόρων οργάνων. Επίσης υπογραμμίζω ότι στα μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε έναν ε, τρίλογο για τον προϋπολογισμό και δεν θα πρέπει να τον αγνοήσουμε για να δοθεί και ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση αυτού του γραφείου. Η Φρανσουάς Κόντ, όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε ποιοι ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Ζανίν Χάνης Πλέσσερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομη και θα σταθώ στο σημείο που μας ανέφερε η συγγήτρια το Κοινοβούλιο όπως και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε μια γρήγορη επίλυση αυτού του προβλήματος και στη γρήγορη δημιουργία αυτού του οργανισμού. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε τίμημα. Ο ρόλος των συμβουλευτικών οργάνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όπως επίσης και η οργάνωση των ε, σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Βέβαια για το θέμα της αλληλεγγύης πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει ένα βήμα προς τα και για το κοινοβούλιο δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στο να προχωρήσει γρήγορα στο να ορίσει τους διευθυντές κλπ. Χρειάζεται ένας ετήσιος όμως απολογισμός στο Κοινοβούλιο και για τα θέματα αλληλεγγύης. Κατανοώ αυτά που λέει η συγγήτρια. Το Συμβούλιο θέλει ένα εκούσιο σύστημα αλληλεγγύης. Εγώ είχα ήδη αρκετές επαφές με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν και έχω πει πολλές φορές ότι το σύστημα δεν δουλεύει ακριβώς γιατί λείπει η ελληνική. Εμείς είχαμε μιλήσει για το 2010 ως οριακή ημερομηνία και έχουμε φτάσει στο 2012. Η ελληνική λοιπόν είναι ουσιαστικότατη. Πώς το Συμβούλιο όμως μπορεί να κάνει κάτι ούτως ώστε και οι 27 να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Όλοι θα πρέπει να δράσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν αλληλεγγύη, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πρέπει να δούμε και πώς προσεγγίζει τα πράγματα το Συμβούλιο. Στην πράξη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη. γιατί στην πράξη τελικά βλέπουμε πολύ συχνά ότι παραβιάζουν οι υπεύθυνοι την αρχή της αλληλεγγύης, μόνο ότι αυτή μπορεί θεωρητικά να έχει αποφασιστεί σε κάποιο αρχικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι από τα κράτη-μέλη λείπει ακριβώ αυτή η αλληλεγγύη. Και φοβάμαι ότι αυτό ενδεχομένω να υπονομεύσει την, το όλο εγχείρημα. Αν δεν εξασφαλίσουμε λοιπόν την αλληλεγγύη, τότε δεν υπάρχει λόγο να δώσουμε καμία συνέχεια στο όλο εγχείρημα. Ο κύριο Γιάνγκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μα την κυρία Τζιν Λάμπερτ, για την πολύ καλή παρουσίασή τη και θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο-τρία ζητήματα και να θέσω και ένα ερώτημα. Από ό,τι φαίνεται η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πολύ σημαντική υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όμω πώ θα εφαρμοστεί η κοινοτική πολιτική για το άσυλο στην πράξη. Ποιο θα έχει πρόσβαση σε όλε αυτέ τι πληροφορίε. Τι είδου πληροφορίε θα διαχέουμε θα έχουν πρόσβαση νομικοί, δικηγόροι, οργανισμοί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι προασπίζονται τα δικαιώματα των ε, προσφύγων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα συμβουλευτικό φόρουμ για την ε, κοινωνία των πολιτών. Θεωρώ ότι αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μάλιστα και εκπρόσωπο ε, τη ε, κοινωνία των πολιτών από μη κυβερνητική οργάνωση στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου τη Υπηρεσία, προκειμένου να μπορεί η υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει πιο καλά θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να είναι σε θέση και των πολιτών να συμβουλεύει την υπηρεσία. Και ποιο ακριβώ θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Για παράδειγμα, στα πλαίσια μια δικαστική διαδικασία, ένα δικηγόρο χρειάζεται κάποιε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Αυτή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο, όσον αφορά για παράδειγμα τη χώρα καταγωγή ενό ατόμου. Θα του δοθούν οι πληροφορίε αυτέ ή όχι. Αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Και τέλο, κύριε Πρόεδρε, η έδρα τη υπηρεσία αυτή. Πού θα είναι η έδρα. Το Συμβούλιο μας είπε ότι θα το αποφασίσουν αυτό τα κράτη-μέλη. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό όμως να γνωρίζουμε πού θα είναι η έδρα. Γιατί αν πρόκειται για μια χώρα η οποία υφίσταται πολύ μεγάλη πίεση από μετανάστε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εξελιχθούν εντελώ διαφορετικά από το να δημιουργηθεί ο οργανισμό αυτό και να έχει την έδρα του σε χώρα πιο ουδέτερη. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε λοιπόν πού ακριβώ θα ιδρυθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ντεγιάνγκ, ο κύριο Στράσε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Είναι σαφές για μας ότι αυτά τα οποία εμείς εδώ ως Γραφείο Υποστήριξης ε, αναφέρουμε είναι μόνο η πορεία προς τα εκεί που είναι ο στόχος μας, δηλαδή σε ένα ενιαίο σύστημα χορήγησης ασύλου για όλη την Ευρώπη, για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης θεμάτων ασύλου για όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό κάθε μέσο και εργαλείο πρέπει να υποστηριχθεί, όταν αυτό υποστηρίζει ότι γοργά θα δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία υποστήριξη στο άσυλο. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την ε, Σουηδική Προεδρία και το Συμβούλιο εφέτος να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα το 2009. Πρέπει ο ένας να ανταποκριθεί στα αιτήματα του άλλου. Έχει νόημα και λόγο στο πρώτο βήμα να είναι εθελοντικός ο χαρακτήρας. Εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν. Έχει νόημα να υπάρχει το best practices, οι βέλτιστες πρακτικές. Έχει νόημα η συναπόφαση για το προσωπικό από πλευράς ε, του Κοινοβουλίου. Και έχει νόημα επίσης κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίζεται μια σε τακτά διαστήματα υποβολή εκθέσεων στην Ευρωβουλή. Είναι σημεία που γοργά πρέπει να τα ολοκληρώσουμε και αυτή η υπηρεσία μέχρι τα τέλη του έτους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μα κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπω θα έπρεπε, πιστεύω. Η προηγούμενη ομάδα, μάλλον η ομάδα την οποία εκπροσωπώ από τι κάτω χώρε, δεν συμφωνεί με την προσέγγιση που υιοθετείται στα πλαίσια του κανονισμού αυτού τη πρόταση κανονισμού θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όσον αφορά τον προπολογισμό, δεν συμφωνούμε με, την, ε, τον προπολογισμό όπως ε, έχει καταρτιστεί στα πλαίσια του κανονισμού αυτού και θεωρούμε ότι οι κάτω χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν την εθνική τους αρμοδιότητα για το άσυλο. Δεν θέλουμε κοινοτική αρμοδιότητα για το άσυλο. Κύριος Μωρές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η Τζιν Λάμπερτ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εντοπίζοντα τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στα πλαίσια του Συμβουλίου. Είμαστε σαφώ υπέρ τη πρόταση τη Σουηδική Προεδρία, η οποία μάλιστα μα καλεί να επιταχύνουμε την νομοθετική διαδικασία. Θα πρέπει όμω αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να έχει μια κάποια αξιοπιστία, να μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Και γι' αυτό το λόγο ζητήματα όπως ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή θα πρέπει να διευθετηθούν με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί αυτό θα προσδώσει μεγαλύτερη εξοπιστία στην τελική υπηρεσία που θα προκύψει. Τα ζητήματα αυτά κάθε άλλο παρασήμαντα λοιπόν είναι επίσης. Κάτι ακόμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να κινηθεί ακόμα περισσότερο προς τη δική μας την πλευρά όσον αφορά το ζήτημα της ε, λογοδοσίας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο θα πρέπει να είχαμε φτάσει όσον αφορά το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Το Συμβουλευτικό Φόρουμ δεν έχει να κάνει μόνο με την εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανισμών. Αναφερόμαστε εδώ πέρα και σε ε, τοπικές αρχές που θα πρέπει και αυτές να εμπλακούν περισσότερο και θα πρέπει να συμβάλλουν. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή ακόμα στην δημιουργία του συμβουλευτικού αυτού φόρουμ, το οποίο θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί με βάση τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί. Σαφώ υπάρχει πολύ καλή πρόθεση από την Προεδρία για να επιληθούν κάποια από τα ζητήματα αυτά και η Τζιν Λάμπερτ έχει εντοπίσει τα τέσσερα αυτά πέντε σημεία τα οποία μα θέλουμε να επιληθούν, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε τελικά μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο που θα έχει αξιοπιστία, που θα διακρίνεται από αξιοπιστία. Το βασικό ζήτημα δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η αξιοπιστία, θα έλεγα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον προλαλή σα, τον προλαλήσαντα, με συγχωρείτε, και να συμφωνήσω, να συγχαρώ την κυρία Τζιν Λάμπερτ, να πω και εγώ ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε γρήγορα και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε όλες τις πλευρές προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε συμφωνία πριν το τέλος του έτους. Είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτό το χειρό μήνυμα ότι κάνουμε κάτι συγκεκριμένο για το ζήτημα αυτό και ότι θα καταφέρουμε τελικά να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξη για το άστιλο. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Όσον αφορά τα κρεμή ζητήματα, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι τα περισσότερα από τα ζητήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα οποία πιέζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι τόσο δύσκολα στη τελευταία ανάλυση. Όσον αφορά την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπηρεσία αυτή, δεν νομίζω τα πράγματα είναι τόσο δραματικά. Τα όσα ζητούμε αυτή τη στιγμή ισχύουν ήδη και για άλλε υπηρεσίε με τι οποίε συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω λοιπόν θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια ειδική συμφωνία στο σημείο αυτό. Θα ήθελα απλώ να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να, από το Συμβούλιο με συγχωρείτε, να έρθει πιο κοντά στη θέση την οποία πρεσβεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το ζήτημα τη αλληλεγγύη. Αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο μας κάνει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με το ζήτημα της αλληλεγγύης και μάλιστα θα έλεγα ότι θα δοκιμάσει και τα όρια της αρχής αλληλεγγύης, στα ζητήματα μετανάστευσης. Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Μπαρό την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι για τα πιλωτικά σχέδια τα οποία έχουν προταθεί στα πλαίσια της Μάλτας, έξι χώρες από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδήλωσαν ενδιαφέρον προκειμένου να επιδείξουν αλληλεγγύη στον τομέα αυτό. Αναφέρομαι, αγαπητοί συνάδελφοι, σε έξι μόνο χώρε από τι 27 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρεται λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα. Ποια είναι τα πραγματικά όρια τη αλληλεγγύη και μήπω θα έπρεπε να επιβάλλουμε μια κάποια υποχρεωτική, δεσμευτική αλληλεγγύη σε σχέση με την εθελούσια αλληλεγγύη που ισχύει αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διακρίνεται σε υποχρεωτική ή προαιρετική, γιατί η αλληλεγγύη είναι αλληλεγγύη, τελεία και παύλα, και απλώς θα πρέπει να υφίσταται, θα πρέπει να υπάρχει. Αυτό που βλέπουμε όμως στην πράξη δεν ανταποκρίνεται στο ευκταίο, σε αυτό το οποίο θα αποκαλούσαμε πραγματικά αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να δώσω βέβαια απάντηση στο ερώτημα αυτό το οποίο θέτω. Πρόκειται όμως για ένα ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντί να δίνουμε ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία στο ζήτημα της εθελούσιας ελεγγύης σε αντιπαράθεση με την ε, υποχρεωτική ελεγγύη ή το αντίστροφο, αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο κύριε Πρόεδρε είναι μια πραγματική αλληλεγγύη η οποία θα εφίσταται στην πράξη και δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το έχουμε εξασφαλίσει ακόμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουζουτήλ και ο κύριος Διαντεμέρα στο τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι η έκθεση βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά χέρια διότι η Τζιν Λάμπερτ ήδη έχει τεράστια εμπειρία στα θέματα ασύλου. Πρόκειται για άτομο το οποίο έχει στρατευθεί στα θέματα ασύλου. Τώρα θέλω να επαναλάβω μια ιδέα την οποία την έχω πει και ξαναπεί πολλές φορές και θέλω να την ακούσει το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Εσύ μίλησες, ε, Τζιν, ε, για το Συμβουλευτικό Φόρουμ, ε, για τη διάρθρωση του, για το Κοινοβούλιο και συμφωνώ μαζί σου που θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να αποφασίζει αλλά και να προχωρήσει ακρόαση του διευθυντή. Αλλά κανένας όμως δεν είπε τίποτα γι' αυτό που είναι και το πιο σημαντικό και είναι η χρηματοδότηση. Το είπε μόνο η Κομισιόν πολύ δειλά στο τέλος. Λοιπόν, θα λειτουργεί αυτό το γραφείο με δανειζόμενο χρήματα από το Ταμείο Προσφύγων. Εντάξει αυτό είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης αλλά δεν θα πρέπει να παραμείνει έτσι η η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα. Δεν μπορούμε εμείς να υποκαθιστούμε την αλληλεγγύη με γραφειοκρατία. Τζιν, αν θέλεις να λάβεις υπόψη σου αυτό το οποίο λέω, σε παρακαλώ να κάνεις κάποια τροπολογία που να αναφέρεται στη χρηματοδότηση. Διότι η Κομισιόν είπε για τη χρηματοδότηση, βέγα, θα δούμε». Λοιπόν, πρέπει να ορίσουμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε αναπτύσσουμε την υπηρεσία αυτή χωρίς να επιβαρύνουμε το Ταμείο Προσφύγων. Λοιπόν, ε, σε παρακαλώ, αν το λάβεις υπόψη σου, να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι καταρχήν σύμφωνος, αλλιώς θα υποβάλω κι εγώ επικοδομητικά μια τροπολογία. έχοντας ακούσει τις απόψεις των μελών που έλαβαν τον λόγο και παρενέβησαν, ίσως για αντιδράσεις και όλα θα μπορούσαμε να ακούσουμε από την εισηγήτρια κυρία Λαμπέρ κάποιες ε, τοποθετήσεις. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ σε όλους εκείνους που συνεισέφεραν με παρατηρήσεις, σχόλια. Θα έπρεπε να καλωσορίσουμε το επικοδομητικό πνεύμα θα έλεγα του Συμβουλίου για το θέμα αυτό και έτσι με επικοδομητικές τροπολογίες σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου να δώσουμε συνέχεια. Αναφέρθηκε στις αρχές της συζήτησης ότι τα κράτη-μέλη έλαβαν μια απόφαση. Θέλουν να υπάρξει η υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο για να υποστηριχθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου που έχουμε ήδη. Τώρα, μέρος του προβλήματος και του θέματος είναι ότι έχουμε τρέχουσες παρεκκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα στο εκτελεστικό, στο επίπεδο εφαρμογών. Και αυτό ανησυχεί κάποιους όταν έχουμε θέματα αλληλεγγύης. Σίγουρα λοιπόν η υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο θα, έχει, θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση και αναβαθμισμένης ποιότητας και σύγκλησης σίγουρα που έτσι θα επικουρεί και θα ε, ολοκληρώνει την αλληλεγγύη. Για συγκεκριμένες παρατηρήσεις και θέματα που εθίγησαν το θέμα για την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα σχετικά. Πώς έχει. Αυτό που συμφωνήσαμε στην Ευρωβουλή δεν πήγαμε πιο πέρα. Είπαμε ότι αυτό θα ήταν υπό τις διατάξεις για την πρόσβαση σε έγγραφα και όσα ισχύουν ήδη και όσα έχει εργαστεί επ' αυτόν το Κοινοβούλιο και έχει εγκρίνει. Αλλά επίσης εξετάζουμε το θέμα αναβαθμισμένης ποιότητας όσον αφορά τα στοιχεία από την χώρα προέλευσης και από κάποιες πιο διευρυμένες πηγές όπως αυτές που εκμεταλλεύονται και παίρνουν πληροφορίες από αυτές τα κράτη-μέλη για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Μια και η αρχική πρόταση ήταν να έχουμε έναν εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών στο εκτελεστικό συμβούλιο, υπήρξε η παναχώρηση από αυτή την αρχική θέση. Μέρος, ο λόγος που συνέβη αυτό εν μέρη είναι ότι υπήρχαν ήδη θα έλεγα ε, θέσεις αμετακίνητες σε σχέση με το συμβουλευτικό φόρουμ και ότι θα έπρεπε να είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του, θα έπρεπε να συνέρχεται σε τακτά διαστήματα και να προσφέρει από την πραγματογνωμοσύνη του. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Υπό τους όρους για τη χρηματοδότηση, υπό τις παρατηρήσεις του κ. Διευτεμέρα, είναι θέμα το οποίο σίγουρα έχει δίκιο επ' αυτού και θα πρέπει να το ξαναδούμε υπό τους όρους της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης πιο μακροπρόθεσμα υπ' αυτών των θεμάτων. Είναι όμως επίσης σαφές από όλα αυτά που ακούσαμε από τα περισσότερα μέλη το σήμερα το απόγευμα είναι ότι θέλουμε να υπάρξει κινητοποίηση και κίνηση για την εμπλοκή και συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Δεν είναι τίποτα που εκπλήσει αυτό, αλλά είναι ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξη για το άσυλο. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι διακυβερνητική υπηρεσία υποστήριξη για το άσυλο. Ο ρόλο λοιπόν είναι προφανέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι καθίσταται σημαντικό. Πρέπει σίγουρα να βρούμε, να εξεύρουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα διέπει τι αρχέ και τι διεργασίε για την παροχή αποτελεσματική και αυθεντική αλληλεγγύη. Αυτά που θα μα πει το Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την απόφαση που θα λάβει η Ευρωβουλή μα. Κάποιε άλλε παρατηρήσει έγιναν. Σίγουρα θα επανέλθουμε στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο επ' αυτών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές για την προσέγγιση που υιοθετήθηκαν και προφανώς θα λάβουμε υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις περαιτέρω διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Any Σας ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για τις πολύ επικοδομητικές αυτές παρατηρήσεις. Πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχουν ε, πολλοί ευρωβουλευτές που έχουν μελετήσει με πολύ μεγάλη προσοχή το όλο ζήτημα. Δύο σύντομες παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, όσον αφορά το ζήτημα της πληροφόρησης. Έχει υποβληθεί μία τροπολογία στα πλαίσια της Κορεπέρ, την οποία θα πρέπει νομίζω να εξετάσουμε, για το άρθρο 11. Δεν προβλέπονται εδώ πέρα προσωπικά δεδομένα και το άρθρο 11 καλύπτει το ζήτημα αυτό όσον αφορά τώρα το ζήτημα της αλληλεγγύης. Πάρα πολλοί ευρωβουλευτέ αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί τρόποι όπου θα μπορούσαμε να πετύχουμε αλληλεγγύη σε κοινοτικό επίπεδο. Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων σίγουρα πρώτα απ' όλα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μέσο το οποίο προωθεί την αλληλεγγύη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταφέρουμε μέσω πιστεύω του Ταμείου αυτού να αυξήσουμε τα πρότυπα αλληλεγγύης. Επίσης, το ζήτημα της επανακατανομής κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων θα πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει. Δεν θα πρέπει να γίνεται συστηματική ανακατανομή, με συγχωρείτε αυτή, ενδεχομένως να λειτουργήσει αρνητικά, να λειτουργήσει σαν μπούμεραγκ και να μην αποτελέσει λύση στο πρόβλημα. Και τέλος, να υπογραμμίσω την στάση της ε, Προεδρίας λέγοντας ότι ε, η πρωτοβουλία αυτή δεν ανήκει απόλυτα στα πλαίσια του υπόλοιπου νομοθετικού πακέτου για το άσυλο, γιατί πρόκειται για έναν κανονισμό που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια υπηρεσία και αν στόχος μας είναι να επιτύχουμε καλύτερη εναρμόνιση, πραγματικά μέσω τη δημιουργία μια τέτοια υπηρεσία θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αρμόνιση σε πρακτικό επίπεδο. Θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε δηλαδή στην πράξη μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Άλλε παρατηρήσει, παρακαλώ, ε, εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανεί. Καμία παρατήρηση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε το ζήτημα αυτό όσον αφορά λοιπόν τη δεύτερη ανάγνωση για το σημαντικότατο αυτό ζήτημα, ζήτημα προτεραιότητας όπως γνωρίζουμε για τη Σουηδική Προεδρία. Ο πρώτος άτυπος τριμερής διάλογος θα γίνει την 1η Οκτωβρίου. Και είμαι σίγουρος ότι θα καταβληθούν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να καταλήξουμε σε κοινή θέση όλα τα εμπλεκόμενα δηλαδή θεσμικά όργανα θα συνεισφέρουν για να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας πάμε στο επόμενο σημείο της σημερίσιας διάταξης, το υπαριθμό 5 και έχει να κάνει με την δημιουργία ενός δικτύου αξιωματικών συνδέσμων για ζητήματα μετανάστευσης. Γνωρίζουμε ότι εδώ πέρα έχουμε μία πρόταση κανονισμού την οποία και θα συζητήσουμε και η οποία τραποποιεί έναν κανονισμό του Συμβουλίου που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2004. Την εποχή εκείνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συμμετάσχει στη διαδικασία διαβούλευσης και είχε γνωμοδοτήσει και πρόκειται για έναν τομέα όπου με απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2004 η διαδικασία της συναπόφασης εφαρμόζεται πλέον. Επομένως, η προτινόμενη τροποποίηση του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να διερευνήσει καλύτερα τις ε, δυνατότητες που θα μπορούσαν να, καλυφθούν μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου εξωματικών συνδέσεων μετανάστευσης και την καλύτερη συνεργασία με την υπηρεσία Frontex. Δεδομένης λοιπόν της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν πρόκειται για πρωτοβουλία, σας υπενθυμίζω, των κρατών μελών, θα ήταν καλό, πιστεύω, να δώσουμε καταρχάς το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στους ε, εκπροσώπους της Προεδρίας Συμβουλίου προκειμένου να μας ενημερώσουν για το πώς έχουν τα πράγματα με την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντίαθ Δεμέρα ο οποίος θα μας ε, παρουσιάσει τις δικές του παρατηρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Ευρωβουλής κυρίες και κύριοι, ο στόχος της πρότασης είναι να προσαρμοστεί αυτός ο κανονισμός υπό το φως της πρακτικής πείρας και εμπειρίας σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο από τότε που η πρόταση υιοθετήθηκε για την δημιουργία νομικής βάσης και τη συνεργασία σε σχέση με την Frontex και τους αξιωματούχους διαμεσολαβητές μεσολαβούντες από πλευρά των κρατών μελών για τα θέματα μετανάστευσης εκμεταλλευόμενη την πείρα τους και εξορθολογώντας σε ένα ορθολογικό πλαίσιο τις διαδικασίες και διασφαλίζοντας επίσης ότι ως συνομοθέτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται με το τακτό και τακτικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίες αυτές οι αλλαγές σε σχέση με αυτή την προώθηση της συνεργασίας μέσα από αυτό το σημαντικό εργαλείο στη συνεργασία σε σχέση με τα όσα υιοθετήθηκαν τον, το 2004 σύνδεσμοι σημαίνει αξιωματούχοι, ε, σύνδεσμοι αξιωματούχοι θα είναι από πλευρά των κρατών μελών εκείνοι που θα δημιουργήσουν αυτή την επαφή και το δίκτυο επαφών σε σχέση με τη χώρα υποδοχής, ώστε να υπάρξει καταπολέμηση και πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των υπηκών τρίτων χωρών όσον αφορά μια απόφαση αποπομπής τους και αυτά ε, εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο και των προξενικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών ή άλλων οργάνων ή θα μπορούσαν και σε σχέση με τρίτε αρχέ και διεθνή θεσμικά όργανα να έχουν επαφές. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφέρω αυτές τι εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο και την πρακτική πείρα που ε, οδηγεί στο να χρειάζεται προσαρμογή αυτή η οδηγία για τη διαχείριση των ε, θεμάτων ε, μετανάστευσης ICONET που άρχισε να λειτουργεί με απόφαση του Συμβουλίου Μάρτιο 2005 για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, παράνομη είσοδο και παράνομη διαμονή σε μια χώρα. Και για την χρήση αυτού του δικτύου εκτίθενται τα σχετικά από την απόφαση της Επιτροπής. Η επιστολή αναφέρει ρητά τι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με το ICONET δεν θα συμπεριλαμβάνει προσωπικά δεδομένα της προσωπικής ζωής ή απόρριτα άλλα στοιχεία τα οποία ε, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται άλλα μέσα για την ε, επικοινωνία σε σχέση με τους ε, υπεύθυνους επιτόπου και για την ανταλλαγή με άλλα κράτη-μέλη είναι στοιχεία κλειδιά για μια διευρυμένη συνεργασία για θέματα μετανάστευσης. Γι' αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαχθεί η χρήση εύκολα προσβάσιμων και προσπελάσιμων εργαλείων σε σχέση με τη μετανάστευση όπως και το ICONET μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού θα διασφάλιζε ότι χωρίς καθυστέρηση θα μπορούσαν να ενημερώνονται οι αρμόδιοι για την περιοχή, την, ε, ένα οργανισμό ή ε, θέματα μετανάστευσης άμεσα. Θα μπορούσε μια συνεργασία να υφίσταται σε σχέση με αυτά τα θέματα με το εμπλεκόμενο κράτος. Έτσι, οι αξιωματούχοι σύνδεσμοι θα μπορούσαν να διαφυλάσσουν τα ε, συμφέροντα ενός και περισσότερων κρατών μελών. Αυτό το οποίο προαναφέρθηκε από τον Πρόεδρο θεσπίστηκε τον Οκτώβριο 2004 και άρχισε να λειτουργεί το 2005, ένα έτος μετά. Μεταξύ άλλων, η Frontex πρέπει να κάνει αναλύσεις κινδύνου. Αυτές οι αναλύσεις κινδύνου πρέπει να βασίζονται στις ε, στα ευρύτερα θεμέλια διαθέσιμων δεδομένων και θα πρέπει να διατίθενται και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Για να υλοποιήσει την αποστολή της η Frontex πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία, λειτουργική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών και η ίδια η Frontex μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνεί οργανισμούς οι αξιωματούχοι αυτοί σύνδεσμοι μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων. Ακόμα δεν, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το δυναμικό από πλευράς Frontex επαρκώς δεσμούς δηλαδή μεταξύ των αξιωματικών συνδέσμων και της Frontex. Έτσι μέσα στο πλαίσιο τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα, διευκολυνθεί η πρόσβαση των ε, υπαλλήλων της Frontex και των επαφών του ε, με άλλους, ε, άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμού. Θα μπορεί να αναλαμβάνεται η πρωτοβουλία να υπάρχουν συναντήσεις σε τακτά διαστήματα μεταξύ των αξιωματικών συνδέσμων και της Frontex. Έχει αρχίσει η συνεργασία όσον αφορά τις οδούς μεταναστευση, migration routes, ταυτοποιώντας τη, τη διαφορετική πορεία εκάστοτε και έχοντας και μια κοινή πλατφόρμα για τους αξιωματούχους για θέματα μετανάστευσης ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα ώστε οι, πιο, οι περισσότερο ενδιαφερόμενοι και με μεγαλύτερη πρωτοβουλία να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο. Όσον αφορά τα καθήκοντα της αρμοδιότητες απαιτείται να συντάσσονται εκθέσεις όσον αφορά την ενισχύη κατάσταση σε κάθε τρίτη χώρα όπου υπάρχουν εκεί σε αυτήν αξιωματούχοι σύνδεσμοι για θέματα μετανάστευσης μια και αυτή τη στιγμή βρίσκονται τέτοιου είδου αξιωματούχοι σε πάνω από 130 χώρε, αυτέ οι διατάξει για την υποβολή εκθέσεων δεν είναι εφικτέ και δεν είναι δυνατόν να ε, ξεπεράσουμε τι ε, ε, την ανάγκη αυτή. Και γι' αυτό θα πρέπει σε τακτά διαστήματα σε συγκε... για συγκεκριμένε χώρε ή συγκεκριμένε ζώνε και χώρε ενδιαφέροντο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλλονται τέτοιε εκθέσει. Όχι μόνο στο Συμβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταχύτατα θα καταλήξουν στη σύναψη μια συμφωνία επί τη προτάσεώ μα και θα μπορέσει έτσι αυτό να προσαρμοστεί και να προαχθεί όπω πρέπει. Ευχαριστώ σα. Ευχαριστώ κύριε Ντόμο. Τώρα εξ της του Συμβουλίου. Η κυρία, η Πέρσον παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θέλω μόνο σύντομα να σας αναφέρω το πώς έχουν επικαιροποιημένα τα πράγματα αυτά σε σχέση με το Συμβούλιο. Στις 23 Σεπτεμβρίου συνήλθε η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τους συνοριακούς ελέγχους. Συζήτησε αυτή την πρόταση σε μια πρώτη φάση τότε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην συνάντησή της ε, υπέβαλε την πρότασή της. Η ομάδα εργασίας συζήτησε το σύνολο της πρότασης, ε, τους τίτλους, ε, το προήμιο, καταδείχθηκε ότι υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία για την υποστήριξη από πλευρά των κρατών μελών υπέρ αυτή τη πρόταση. Η ομάδα επικεντρώθηκε σε δύο ελάσσο ίσονο σημασία τροπολογίε ή τροποποιήσει, μάλλον γλωσσική φύσεω παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. Δεν αλλάζουν τίποτα επί τη ουσία αυτέ οι γλωσσικέ προσαρμογέ. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση, για μια πολύ καλή στην πρακτική εφαρμογή και στην εκτέλεσή τη πρόταση και καταδείχθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια 30 λεπτών ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία. Πιο γοργά δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Η υποστήριξη ήταν πραγματικά συντριπτική λοιπόν και δεν ε, ήταν περίπλοκο, καθόλου σύνθετο ή περίπλοκο το θέμα ώστε να καθυστερήσουμε. Γι' αυτό η Προεδρία θα ήθελε αυτή η πρόταση να προαχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και αν η συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα στο Συμβούλιο εξελιχθεί με τον ίδιο ταχύ τρόπο και τις ίδιες ταχύες διεργασίες, τότε μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στο Συμβούλιο θα μπορέσουμε να λάβουμε θετική απόφαση σχετικά. Αλλά φυσικά θα θέλαμε να έχουμε και τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου τις οποίες θέλουμε να λάβουμε υπόψη, να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση με άλλα λόγια με την Ευρωβουλή. Και γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι φυσικά να αφιερώσουμε τον αναγκαίο χρόνο για το Ευρωκοινοβούλιο να εισακουστούν οι απόψεις του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πέσον. Και τώρα ας ακούσουμε από πλευράς του κυρίου μέρα για την πρώτη ανάγνωση της έκθεσης στα σχετικά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή την αναλυτικότατη παρουσίαση της Κομισιόν με την οποία συμφωνώ ουσιαστικά. Και σήμερα το πρωί συνεδρίασα με τη Μαριάν Πέρσον και τους ε, συνεργάτες της για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ακριβή θέση του Συμβουλίου σχετικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι πρόκειται για μία έκθεση συναπόφασης. Πρόκειται για μία πρόταση απλή με λίγες τροπολογίες. Απλές τροπολογίες. Επιτρέψτε μου λοιπόν πρόεδρε να σας πω ότι αφού κάνω εγώ την παρουσίασή μου και ακούσουμε και τους συναδέλφους να σας διατυπώσω και το χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να μπορέσει να εγκριθεί η έκθεση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Θέλω να πω ότι τελικά στην Σεβίλη και στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ρίζα αυτής της έκθεσης, διότι εκεί για πρώτη φορά ε, καθοριστικά προωθήσαμε την δημιουργία αυτών των αξιωματούχων. Και όλη αυτή η πρόταση ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να κουράσω τους συναδέλφους, γιατί έχουμε ιδιαίτερα φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Εμείς αυτό που θέλουμε με αυτή την έκθεση είναι να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε το ρόλο όλων αυτών των αξιωματούχων και να απορροφήσουμε όλες αυτές, όλο αυτό το δυναμικό μέσα στο Frontex. Δηλαδή, οι, σύνδεσ... υπάλληλοι των συνδέσμων μετανάστευσης ε, και του Frontex να γίνουν ουσιαστικά ένα. Δημιουργία λοιπόν δικτύων και όσον αφορά στο σύστημα πληροφορικής δεν επιτρέπεται να γίνεται διαβίβαση προσωπικών στοιχείων. Θα μου πείτε άμα δεν μπορούμε εμείς να διαβιβάσουμε προσωπικά στοιχεία τότε σε τι συνίσταται η ανταλλαγή στοιχείων. Συνίσταται στο να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας τις διάφορες ροές μεταναστών, τα στοιχεία του δουλεμπορίου, το modus operandi, τον τρόπο λειτουργίας δηλαδή των κυκλωμάτων το πώς ε, γίνεται η πλαστογραφία των διαβατηρίων και λοιπά και λοιπά λέει ο μιλητής πιστεύω λοιπόν ότι αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο ποιοτικά ανώδυνες είναι οι τροπολογίες ε, του Συμβουλίου που είναι καθαρά ε, ε, ψηλοπράγματα του τύπου ας πούμε προτείνουν το θα πρέπει να αντικατασταθεί με το θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία και για τη νομική βάση που είναι το άρθρο 63.3 και το 66 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Όπως επίσης και η βάση του 363 κανονισμού του 2004. Λοιπόν, στο τέλος κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να δώσω και χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, ζήτησαν το λόγο η κυρία Χένις Πλέσσερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και με προφορικές ερωτήσεις εγώ είχα ζητήσει να μου διευκρινίσουν αυτό το θέμα των αξιωματικών και μου είχαν πει πολλές φορές, μου είχαν απαντήσει ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ήταν στην διάθεση του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για την υποβολή των διαφόρων εκθέσεων. Λοιπόν, μου φαίνεται, δεν είμαι όμως σίγουρη και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε, ότι έχει λυθεί πλέον το θέμα και υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις. Τώρα, όταν πρόκειται για τις επιβιβάσεις σε αεροπλάνα. Υπήρχε ένα πρόβλημα της ε, Κομισιόν σχετικά με την αποδοχή των διαφόρων κανόνων και προδιαγραφών που επιτρέπουν την επιβίβαση στα αεροπλάνα. Θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν αν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλε. Συμφωνώ με το ζήτημα αυτό, είναι ακόμα ασαφές. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς κάνουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι, τι συζητούν στι συνεδριάσεις που κάνουν και στι οποίε θα κάνουν ακόμα περισσότερο από ό,τι φαίνεται στο μέλλον. Σε μία από τι τροπολογίε για το άρθρο 6 λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει σε τήσια βάση εκθέσεις που θα περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ενδυναμώνεται το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων και το πώς συνεργάζεται τελικά με τους άλλους ηθήνοντες. Αυτό που χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι περισσότερες πληροφορίες ή αιτήσει εκθέσεις για το πόσο καλά χρησιμοποιούν το ίντερνετ ή το ίκονετ πιο συγκεκριμένα οι αξιωματικοί σύνδεσμοι. Αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοι. Και έτσι θα καταφέρουμε να δούμε και αν ε, όντως οι αξιωματικοί σύνδεσμοι καλύπτουν τις ε, εργασίες τις οποίες υποτίθεται ότι θα πρέπει να καλύπτουν ή αν θα πρέπει ουσιαστικά να τους δώσουμε άλλες αρμοδιότητες. Τώρα, στα πλαίσια της εξέτασης του κανονισμού αυτού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις πληροφορίες ακριβώς εκείνες τις οποίες υποτίθεται ότι συλλέγουν οι εξωματικοί σύνδεσμοι. Πληροφορίες που δεν αναφέρονται καθόλου στην πρόταση κανονισμού. Δηλαδή πώς μεταχειρίζονται για παράδειγμα τους μετανάστες ε, στην ε, χώρα προορισμού ε, συγκεκριμένες αρχές. Δεν γνωρίζουμε καθόλου τη μεταχείριση στοιχαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να αναφέρεται γιατί και αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευση σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και τι μεταχείριση τυχαίνουν από τις χώρες στις οποίες φτάνουν. Και δύο πληροφορίες σημαντικές που, μάλλον αυτές είναι δύο σημαντικές πληροφορίες που αποσιάζουν από την ε, νέα αυτή πρόταση καονισμού. Σας ευχαριστούμε. Εκτός μικροφώνου, ο Πρόεδρος. Maybe some additional points from the... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως ή το Συμβούλιο θα ήθελα να προσθέσουν κάτι. Κύριε Ντόμπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω ότι ε, οι εξωματικοί σύνδεσμοι διορίζονται από τις εθνικές αρχές, από τα κράτη-μέλη ουσιαστικά. Δεν εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπροσωπούν ουσιαστικά το κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται. Και ο κανονισμός προβλέπει μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους εξωματικούς συνδέσμους. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως επιθυμεί να πάρει το λόγο. Κυρία Πέρσον. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φυσικά ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών και τα σχόλιά τους και σίγουρα θα ενημερώσουμε για την περαιτέρω συνάντηση στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο κύριε presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχόλια της Ζωνίν και της ε, συναδέλφου μας για, τους, ε, για το τι πράττουν οι αξιωματικοί συνδεσμοί. Μα αυτό λέγεται στον κανονισμό 334. Τι κάνουν λοιπόν. Συμβάλλουν στην ε, πρόληψη και καταπολέμηση της ε, λαθρομετανάστευσης, στην διαχείριση της ε, λαθρομετανάστευσης, τον επαναπατρισμό κλπ. Αυτά λέει ο κανονισμός. Αυτό που εμείς ε, τώρα θέλουμε να κάνουμε με αυτήν την νομοθετική πράξη είναι να τροποποιήσουμε τα άρθρα 3, 4 και 6 αυτού του κανονισμού. Εγώ δεσμεύομαι ιδιαίτερα να λάβω υπόψη μου τις προτάσεις των συναδέλφων. Θα ήθελα τώρα, Πρόεδρε, να προτείνω το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας, γιατί επαναλαμβάνω, πρόκειται για μία έκθεση απλή, δεν υπάρχουν ε, προβλήματα. Το μόνο που κάνει είναι να βελτιώνει τον ήδη υπάρχοντα κανονισμό. Προτείνω λοιπόν, Πρόεδρε, στις 4 ή 5 Νοεμβρίου να έχουμε το έγγραφο εργασίας, μετά να ανοίξει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 6 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι και προτείνω 16 Νοεμβρίου να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας ή στην συνεδρίαση της 1ης ή Δευτέρας Δεκεμβρίου και φυσικά αν υπερψηφιστεί η έκθεση να κατατεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση στις 14 Δεκεμβρίου. Δεν έχω τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντεμέρα. Θα έλεγα λοιπόν έγινε η πρόταση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ήδη. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση μεταξύ των μελών της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής υιοθετείται. Θα λάβουμε υπόψη ακριβώς αυτή την πρόταση ώστε να είναι συμβατή και να συνάδει με την ημερήσια διάταξη και τις εργασίες των άλλων κοινοβουλευτικών σωμάτων και φορέων, ιδιαίτερα με τις εργασίες Ολομέλειας. Αν συμφωνείτε λοιπόν τώρα, νομίζω ότι αυτό το σημείο συζητήθηκε και είναι έτοιμο το χαρτοφυλάκιο να δοθεί συνέχεια σε αυτό, να προωθηθεί. Και στα επόμενα σημεία περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε? Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τώρα τα σημεία 6 έως 11. Διότι όλα αυτά τα σημεία από κοινού αφορούν εκθέσεις ε, που έχει αναλάβει να συντάξει ο κύριος Μπουσούτιλ. Θα πρότεινα λοιπόν, σαν συνέπεια τούτου, να έχουμε μια κοινή συζήτηση. Κοινή συζήτηση από το σημείο 6 ως το 11 των συναφών αυτών θεμάτων. Το 6 αφορά συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου σε σχέση με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίου για σύντομη διαμονή. Το 7 το ίδιο για τον Μπαρμπάντος για σύντομη βραχία διαμονή. Το 8 για την ε, Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου Σεντ Κίτς ε, και Νέβης για διαμονή. Το σημείο 9. Απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μπαχάμας, των νησιών Μπαχάμες. Και το ίδιο το 10 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγουας και Μπαρμπούντα όσον αφορά την απαλλαγή υποχρεώσεων θεωρήσεων διαβατηρίων. 11 για τις Σεϊχέλες πάλι το ίδιο, απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων για βραχία διαμονή. Όλα αυτά τα σημεία, δεν κάνω λάθο λοιπόν, είχαν, τα είχε αναλάβει ο κύριος Μπουσούτιλ ως εισηγητής αρμόδιος για την παρουσίαση των σχολείων και παρατηρήσεων του. Έχει τον λόγο λοιπόν να μας παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. Ο κύριος Μπουσούτη, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Λιγότερο χρόνο θα χρησιμοποιήσω, θα αναλώσω από ότι εσείς εισάγοντας όλες αυτές τις εκθέσεις, διότι είναι απλές και εύληπτες αυτές οι εκθέσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπόρεσα να επισκεφθώ και αυτό με θλίβει βέβαια αυτές τις χώρε. Πάντα θα ήθελα και πολύ θα ήθελα να τις έχω επισκεφθεί. Είναι πολύ σύντομε λοιπόν αυτές οι εκθέσεις όπως είπα και αφορούν το χωρί θεωρήσει διαβατηρίων ταξίδι των υπηκών αυτών των χωρών στην ευρωπαϊκή κοινότητα και των πολιτών τρίτων χωρών που αναφέρατε κύριε Πρόεδρε για μέγιστη περίοδο τριών μηνών για βραχία διαμονή. Το κύριο θέμα σε αυτές τις εκθέσεις λοιπόν και θα έλεγα κιόλας και το μόνο ζήτημα που υφίσταται σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις αφορά την αρχή της αμοιβαιότητας. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό. Εμείς έχουμε εδώ μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία εμείς παρέχουμε αυτό το οποίο μας παρέχουν και οι άλλοι από την άλλη όχθη και οι πίκοοι αυτών των τρίτων κρατών έχουν αυτά τα οποία τους δίνουμε εμείς αλλά έχουμε και εμείς τα ίδια δικαιώματα. Δηλαδή η αρχή της αμοιβαιότητας υπάρχει της αμοιβαίας αυτής ανταπόδοσης είναι σεβαστή. Κατανοώ ότι ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι παρόν εδώ, είναι πα... Ε, τη συνάντησα εχθές για να συζητήσω αυτό το θέμα μαζί της. Πιστεύω ότι πραγματικά θα έπρεπε να παρέμβει εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσει μια διασφάλιση, μια επιβεβαίωση για το θέμα αυτής της αμοιβαιότητας που θα ισχύει όσον αφορά το εγχείρημα αυτό της ε, απαλλαγής υποχρέωσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες αυτούς. Και όταν θα έχει διασφαλιστεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, τότε προτείνω αμέσως να υπερψηφίσουμε, να ψηφίσουμε για την έγκριση αυτών των εκθέσεων αύριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουσούτη για την σαφήνεια και συντομία της παρουσίασής σας. Με ενημέρωσαν ότι ο εισηγητής δεν έχει την πρόθεση να καταθέσει τροπολογίες και έτσι λοιπόν προτείνω χάρη αυτής της σαφήνειας να έχουμε την προθεσμία για τροπολογίες για τα μέλη που θέλουν να καταθέσουν κάποια τροπολογία. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σωστό να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει. Και η Προεδρία του Συμβουλίου. Πρώτα, από πλευρά της Προεδρίας του Συμβουλίου, η κυρία Λέιλα Ελφανίδη παρακαλώ θα λάβει τον λόγο από τη Σουηδική Προεδρία. Παρακαλώ. Η κυρία Ελφαλίνη, παρακαλώ. Θα ήταν ε, ε, εδώ ουσιαστικά η άλλη συνάδελφος που θα έπρεπε να παρέμβει. Έχει τον λόγο. Λοιπόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο τι έκανε. Απεφάσισε αυτές οι έξι, τα έξι κρατήδια, στα αποκαλέσω έτσι, να αναβληθεί η προσυπογραφή των ε, απαριθμούμενων σε σχέση με την απαλλαγή δηλαδή χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων. Και αυτό το αναβάλουμε ώστε να υπάρξει η ταυτόχρονη αμοιβαιότητα και αποφασίστηκε αυτή η απαλλαγή να μην ε, συνάπτεται με διμερείς συμφωνίες, να μην ε, έγκυται μέσα σε πλαίσιο ε, διμερών συμφωνιών, αλλά σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας. Τον Ιούνιο 2008 το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με αυτά τα κρατήδια προς αυτόν τον στόχο. Οι διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν και τον Νοέμβριο 2008 μπόρεσαν να ε, μονογραφηθούν αυτές οι συμφωνίες. Τον Απρίλιο 2009 έλαβε την απόφαση το Συμβούλιο επ' αυτών των συμφωνιών και τώρα αναμένει το Συμβούλιο μόνο την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε αυτές οι συμφωνίες να μπορέσουν να ε, εφαρμοστούν. Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες σας προς επικύρωση και μόλις θα είναι έτοιμη η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα έχει συνταχθεί αυτό το σημείο θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης του Συμβουλίου, ώστε αυτό, αυτή η συμφωνία το δυνατόν ταχύτερα να μπορέσει να εφαρμοστεί. Thank Σας ευχαριστώ. Και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ντάφνη Γόγκου, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω, θα είμαι σύντομη. Καταρχάς, να στηρίξω τις παρατηρήσεις που έκανε ο εισηγητής. Το βασικό ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε στα πλαίσια της πρώτης συμφωνίας για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα της αμοιβαιότητας και της ασφάλειας δικαίου. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία πρόταση και είπε ότι τα έξι αυτά μικρά κράτη κληρούν όλα τα βασικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν στα πλαίσια του κανονισμού 539 και επομένως μπορούν να περάσουν στον θετικό κατάλογο. Τον Ιανουάριο του 2007 στη συνέχεια ήταν σαφέστατο ότι οι χώρες αυτές πρέπει να αποτελέσουν τμήμα του θετικού καταλόγου του κανονισμού 539 και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρότειναν η θέση σε ισχύ της εξαίρεσης ε, από τον κανονισμό για την υποχρέωση θεώρησης για τις χώρες αυτές θα αρχίσει να ισχύει μετά την ε, εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση και εφαρμογή τη πρώτη συμφωνία για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση, αμέσω δηλαδή μετά. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την κοινή μα πολιτική για τι θεωρήσει, δέκα χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε το πρώτο εγχείρημα μια τέτοια πολιτική. Βρισκόμαστε πλέον λοιπόν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Περνάμε δηλαδή στην ολοκλήρωση, στην υπογραφή μιας συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις χώρες αυτές και συνοδεύεται ο κανονισμός αυτός στη συνέχεια με τις απαραίτητες αυτές ρυθμίσεις προκειμένου να καταφέρουμε να αγγιηθούμε την αμοιβαιότητα για τους πολίτες μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει και αυτοί να χαίρουν του ίδιου καθεστώτος σε σχέση με τις αναφερόμενες τρεις, τρίτες χώρες. Επομένως, οι κανόνες που ισχύουν για τις θεωρήσεις θα είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους κανόνες που προβλέπονται στην Συμφωνία για την Απαλλαγή από την Υποχρέωση Θεώρησης. Δηλαδή προβλέπονται ακριβώς οι ίδιοι κάτοχοι διαβατηρίου, ακριβώς οι ίδιοι δικαιούχοι, Προσπαθούμε λοιπόν για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο προδιαγραφών, ένα μοντέλο διατάξεων όσον αφορά την πρώτη αυτή συμφωνία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση. Θέλουμε ακριβώ να έχουμε όλε αυτέ τι νομοθετικέ εγγυήσει που θα διασφαλίσουν πλήρη αμοιβαιότητα για όλου τους πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες για να σας πω πώς διευθετείτε το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Να σας πω απλώς ότι ε, ορισμένοι θα γνωρίζετε τι συνέβη πρόσφατα όταν ε, ε, ο Καναδάς αποφάσισε να επαναφέρει την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Τσεχίας πολύ σύντομα θα γνωρίσουμε περισσότερο ποια είναι η τοποθέτηση επίσημη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εμιβαιότητα θα καλύπτονται και τα ζητήματα αυτά και θα ζωθεί κατά αυτόν τον τρόπο μια πλήρη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Από πλευρά των Ευρωβουλευτών, ο κύριος Μπρόνς, παρακαλώ. Ενώ είμαι υπέρ της κατάργησης περί της γραφειοκρατίας όσον αφορά τουρίστες αμφωτέρωθεν η κατάργηση θεωρήσεων διαβατηρίων δεν θα ενίσχυε, ας το πούμε έτσι, περαιτέρω παράνομη μετανάστευση αν ε, ξεπερνούσαν την περίοδο διαμονής τους ε, στα κράτη μας ε, εφόσον αυτές οι αρχές ε, θα έχουν θεσπιστεί θα υπάρξουν περαιτέρω προτάσεις ε, για ε, τέτοιες χορηγήσεις απαλλαγών για χορηγήσεις διαβατηρίων για υπηκός μεγαλύτερων χωρών κρατών όπου θα μπορούσαν τα, οι αριθμοί τους να είναι μεγαλύτεροι στην Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράης παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Περίπου 800.000 ε, υπήκοοι Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέπτονται αυτά τα νησιά, αυτά τα κρατήδια. Θέλω να υποστηρίξω απόλυτα τις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Μπουσούτη για την αμοιβαιότητα, για τα πρακτικά. Με εκπλήσει ότι δεν πήγε σε αποστολή διαρευνητική σε αυτά τα κρατήδια, σε αυτά τα νησάκια. Με, με απογοητεύει Σάιμον Μπουσούτη αλλά αυτό το λέω για να απορριφθούν σε σχέση με τις παρατηρήσεις ε, του προηγούμενου προλαλήσαντος. Ε, πρέπει σε ατομική βάση να μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ναι, εσείς παρακαλώ. Euh, euh, Θα είμαι πολύ σύντομη Πέρα από τα μικρά αυτά αστεία που ακούσαμε, θα ήθελα να εξασφαλίσουμε στην πράξη ότι ε, οι πολίτες αυτοί οι οποίοι έρχονται από τις χώρες αυτές θα πρέπει σαφώς να τυχαίνουν ε, ανάλογης υποδοχής εδώ πέρα με αυτή που ελπίζουμε και εμείς να τύχουμε όταν πηγαίνουμε στις χώρες αυτές όσον αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχία διαμονή. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο. Όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό γνωρίζουν ότι θεωρήσεις βραχίας διαμονής αποτελούν ένα ζήτημα φαύλου κύκλου θα έλεγα όλο και περισσότερα πολλές φορές θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα πολλών πολιτών, ιδίως από τις ε, χώρες ε, του Νότου και αυτό επηρεάζει και τις εμπορικές συναλλαγές με τους εμπόρους από τις χώρες αυτές, αλλά και τις ανταλλαγές των σογγικών με τους αθλητές από τις χώρες αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν να, να καταργούμε τις θεωρήσεις αυτές βραχίας διαμονής. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες που θέλουν να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά, αν διατηρούμε το σύστημα υποχρέωση θεώρηση βραχία διαμονή, ουσιαστικά σπρώχνουμε του ανθρώπου αυτού στην παράνομη μετανάστευση. Όσον αφορά το προτινόμενο κείμενο, εμείς είμαστε σαφώ υπέρ του κειμένου αυτού, ε, να έχουμε κάποιες ε, μικρές ανησυχίε Τι εννοείται όταν λέτε έγκυρο διαβατήριο, είναι αρκετά σαφής ο όρος αυτός για μένα από νομική πλευρά. Ευχαριστώ. Mr. Bonds, please. Ο κύριος Ευχαριστώ. Κυρίως οι χώρες της Καραϊβικής είναι χώρες διαμετακόμισης, διέλευσης για ναρκωτικά που παράγονται στην Νότια Αμερική. Μέσω αυτών των κρατηδίων στην Καραϊβική τα ναρκωτικά περνάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διοχετεύονται εκεί ή στη ΣΥΠΑ. Πέρα από αυτό υπάρχει ξέπλυμα χρημάτων σε αυτά τα νησίδια, σε αυτά τα κρατήρια. Γι' αυτό το κόμμα μου είναι κατά της Κατάργηση θεωρήσεων διαβατηρίων σε σχέση με αυτέ τι χώρε και για τι πρόσθετε εγγυήσει που χρειαζόμαστε σε σχέση με την Ολλανδία. Είμαστε κατά τη απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων για αυτέ τι χώρε. Σα ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστηρίζω την θέση του εισηγητή του κυρίου Μπουσούτη όχι θέσει άλλων που ακούστηκαν στη συζήτηση. Όμω, όμως, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είναι σημαντικό υπό το πρίσμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλε οι σχέσει που έχουμε με αυτέ τι χώρε η ελευθερία, ελεύθερη κυκλοφορία και η υπέρβαση αντιμετώπιση γραφειοκρατία, να τι εκμεταλλευτούμε διπλωματικά ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Να εμβολιάσουμε αυτέ τι χώρε δηλαδή έναντι μια πανδημία που είναι πολύ σοβαρότερη από τη γρήπη, που είναι η φορολογική παράδειση. Είναι στο πλαίσιο μια πολύ ευρύτερη πολιτική και εδώ συγκεκριμένα θα πρέπει να δραχτούμε τη ευκαιρία ώστε οι χώρε αυτέ που είναι φίλε χώρε να μπορέσουν μέσω της νομιμότητας ε, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να μην οξυνθούν τα προβλήματα με μια κρίση όπως αυτή που περνάμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και επανερχόμαστε λέει ο Πρόεδρος στον κύριο Μπουσούτιλ. Αν κατάλαβα σωστά, ο εισηγητή μα πρότεινε να εγκριθεί η απόφαση αυτή αύριο στην ψήφισή τη, στην ψηφοφορία. Καλό είναι να υπάρξει μια προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μέχρι τι 6 το απόγευμα, το βράδυ απόψε, 18.00 η ώρα κατάθεση τροπολογιών, η προθεσμία που θα εκπνεύσει τότε. Μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι τότε, αύριο να τις ψηφίσουμε. Κύριε Μπουσούτη, τι λέτε. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συμφωνώντα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που προτείνατε για την κατάθεση τροπολογιών και την ψήφιση αύριο. Όμω επίση να ευχαριστήσω και του Ευρωβουλευτέ, τα μέλη, που συνεισέφεραν για αυτή τη σύντομη αλλά ζωντανή αναζωογονημένη συζήτηση. Να αποσαφηνίσω δύο σημεία. Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που τρίτε χώρε ε, από τον αρνητικό κατάλογο εγγράφονται σε ένα θετικό πίνακα, σε ένα θετικό κατάλογο για θεωρήσει διαβατηρίων. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν το κάνουμε για πρώτη φορά αυτό σε σχέση με τρίτες χώρες. Δεύτερον, θέλω επίσης να αποσαφηνίσω ότι αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, δηλαδή όλους τους κανονικούς πολίτες, εκτός από, εκτός από τον σκοπό ε, άσκησης επαγγέλματος επαμοιβή που τότε η χορήγηση θεωρήσεως απαιτείται μόνο για αυτό το περιορισμένο εύρος, για αυτό το φάσμα. Έτσι λοιπόν νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Άλλα σχόλια από την Προεδρία ίσω παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Ε, euh, Μία διευκρίνηση από την Κομισιόν σχετικά με την εντολή. Εμείς έχουμε εντολή για τη διαπραγμάτευση θεωρήσεων με τη Βραζιλία. Πρόκειται για την ίδια αντίληψη που θέλουμε να αναπτύξουμε με τρίτες χώρες ούτως ώστε η Κομισιόν να έχει την νομική ασφάλεια για την αμοιβαιότητα μεταξύ των, ε, μεταξύ των τρίτων χωρών και των πολιτών μας. Επίσης ένα σχόλιο. Η κατάργηση των θεωρήσεων δεν σημαίνει ότι καταργούνται και οι έλεγχοι στα σύνορα. Δηλαδή όσοι είναι μπλεγμένοι σε, παράνομες, ε, σε, παρα, σε παρανομίες φυσικά και συλλαμβάνονται στα σύνορα. Παραμένουν οι έλεγχοι των εξωτερικών μας σύνορων ούτως ή άλλως. Ε, σχόλιο εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, θα έλεγα Ολοκληρώσαμε με αυτό το σημείο, με αυτά που είπαμε. Εντάξει, προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Και αυτό είναι το σημείο υπαριθμών 12. Είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία. Είναι αυτή μια έκθεση που έχει αναλάβει να συντάξει η κυρία εξέχουσα προσωπικότητα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη. Πρέπει όμως να ε, ζητήσουμε συγγνώμη, απουσιάζει η συγγήτρια, δεν είναι σε θέση για προσωπικούς λόγους λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων να παραστήσει η σημερινή συνάντηση. Ο Αντιπρόεδρος λοιπόν, ο κύριος Τζακολίνο της Επιτροπής μας θα λάβει τον λόγο εξ ονόματός της. Υπενθυμίζω όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα κύριο αίτημα και μέλημα της Επιτροπής μας το θέμα των παιδιών. Είχαμε υιοθετήσει διάφορες εκθέσεις στο παρελθόν για αυτό το θέμα και μια έκθεση από την κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη την άνοιξη κιόλας που είχαμε συστάσεις για το πόσα η Ευρωβουλή θα ήθελε να εκτελεστεί η απόφαση πλαίσιο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και η παιδική πορνογραφία, πώς θα θέλαμε να προσαρμοστεί, να επικαιροποιηθεί. Ακολούθησε αυτή την έκθεση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συζητούμε σήμερα. Έτσι λοιπόν πρώτα και κύριε αυτό που θα κάνουμε είναι θα δώσουμε τον λόγο ε, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά θα παρέμβει η Σουηδική Προεδρία και μετά από τα σχόλια και παρουσίαση αυτών των οργάνων, ο κύριος Τζακολίνο λάβει τον λόγο εξ ονόματο κυρία Αντζελίλη. Ο εκπρόσωπο λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρόν αυτό ή εκείνη. Ναι, εδώ είμαι. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών αποτελεί τμήμα ενός νομοθετικού πακέτου. Συνδυάζεται δηλαδή με την πρόταση για την ε, εμπορία ανθρώπων, ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και οι δύο προτάσεις έχουν μια σφαιρική ολιστική προσέγγιση, πράγμα το οποίο σημαίνει Πέρα από τις διατάξεις που έχουν να κάνουν καθαρά με ποινικό δίκαιο, έχουμε συμπεριλάβει στην πρόταση κάποιες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, με τις έρευνες, τη δίωξη, με την προστασία των θυμάτων. Είμαστε πεπισμένοι ότι η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα το οποίο συζητάμε, δηλαδή όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών και την παιδική πορνογραφία, Και ο γενικό στόχος εδώ πέρα μια νέας νομοθεσία είναι να εξασφαλίσει καλύτερη προστασία των παιδιών, τα οποία πέφτουν θύματα των ιδεχθών αυτών εγκλημάτων. Η πρόταση βασίζεται σε μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και εμπνέεται ουσιαστικά από τη σύμβαση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη σύμβαση Λαντσαρότε, και θέλουμε όμως, ξεκινώντας από τη σύμβαση αυτή, να πάμε ακόμα πιο πέρα. Να μην περιοριστούμε δηλαδή στα όσα λέγονται σε αυτή τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, να βγούμε από τα πλαίσια της σύμβασης αυτής και να προχωρήσουμε πέρα από τη σύμβαση Λαντσερότε. Όσον αφορά τώρα σύντομα για το περιεχόμενο της πρότασης. Καταρχάς, προβλέπεται εδώ πέρα ένα γενικότερο πεδίο εφαρμογή όσον αφορά τις α, περιπτώσεις εκείνες όπου θα ποινικοποιεί τη σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και η παιδική πορνογραφία. Το πεδίο εφαρμογή είναι πιο ευρύ ως προς ε, διάφορα ζητήματα. Καταρχάς, όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση, καλύπτουμε εδώ πέρα όλες τις εγκληματικές ε, δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όσον αφορά την παιδική πορνογραφία, δεν προβλέπεται εδώ μία εξαίρεση, δεν επιτρέπεται καμία εξαίρεση. Και επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τις ε, τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στα πλαίσια της τεχνολογίας, της επικοινωνίας. Δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε κάποια νέα εγκλήματα, όπως το grooming, το να προσελκύει κανείς παιδιά μέσω του ίντερνετ, για παράδειγμα, με στόχο τη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση. Το να προσπαθεί κανείς να δελεάσει δηλαδή ένα παιδί μέσω του ίντερνετ. Ποινικοποιείται δηλαδή και αυτή η δράση αυτή. Δεύτερος στόχος ποινικό αν θέλετε, είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εναρμόνιση των κυρώσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολύ σοβαρά εγκλήματα και επομένως αναμένεται από όλες τις χώρες και ένα υψηλό επίπεδο κυρώσεων κυρώσεις δηλαδή οι οποίες θα είναι ανάλογες ε, τη σοβαρότητα του εγκλήματο. Όσον αφορά τώρα τι διώξει, τι ποινικέ διώξει, προβλέπεται εδώ πέρα μία νέα διάταξη εξ officio, αυτεπάγγελτα δηλαδή, και επίσης έχουμε και κάποιες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ε, χρήση συγκεκριμένων ε, μέσων ερευνών, όπως για παράδειγμα κρυφές μυστικές έρευνες online που θα γίνονται μέσω του διαδικτύου δηλαδή. Το μέσο αυτό, το εργαλείο αυτό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχές σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει χρησιμοποιηθεί. Τώρα, όσον αφορά την δικαιοδοσία, το ζήτημα εδώ πέρα είναι αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο. Προσπαθούμε να πάρουμε ένα μια αποφασιστική, να προωθήσουμε μια αποφασιστική ε, απόφαση. Το ζήτημα είναι δύσκολο, αυτό έχει φανεί και από τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προσπαθούμε εδώ πέρα να καταπολεμήσουμε τον λεγόμενο σεξουαλικό τουρισμό. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ταξιδεύουν στο εξωτερικό προκειμένου να διαπράξουν το έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών σε μια άλλη χώρα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι διαμένοντες μόνιμα ή συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να διώκονται για τέτοια δικήματα τα οποία διαπράττουν στο εξωτερικό ακόμα και αν δεν προβλέπεται η αρχή του double criminality. Επίσης προβλέπονται και πολλές άλλες διατάξεις όπως ε, η μη τιμωρία του ε, θύματος για εγκλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το θύμα, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν περάσει στην πορνεία μέσω της σεξουαλικής όμως εκμετάλλευσης επειδή ουσιαστικά κάποιος έχει σπρώξει προς ε, την, το δρόμο αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά και θα πρέπει τα παιδιά τα οποία έχουν πέσει θύματα να προστατεύονται από την περίπτωση εκείνη που θα πέφτουν εκ νέου θύματα εξαιτίας της ε, καταστολής ε, που προβλέπεται από ένα κράτος μέλος. Δηλαδή, θα πρέπει να προβλέπεται αυτό και στα πλαίσια των και στα των ακρίσεων, να μην προβλέπεται μία επιπλέον τραυματοποίηση των παιδιών. Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Βλέπονται εδώ πέρα διάφορες διατάξεις όσον αφορά την ε, πρόληψη. Καταρχάς, κάποια προγράμματα τα οποία απευθύνονται στους ε, ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν περιπέσει σε τέτοια εγκλήματα ή για τους οποίους υπάρχει υποψία ή οι οποίοι φοβούνται ότι θα μπορούσαν να περιπέσουν σε τέτοια εγκλήματα. Θα πρέπει να προβλέπονται λοιπόν τέτοια προγράμματα πρόληψης τόσο για τους ε, δυνάμει αν θέλετε

τα, τις ιστοσελίδες αυτές, ιδίως όταν έχουν την έδρα τους εντός αγωγικών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να κάνουμε σε μια πρώτη φάση, είναι να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε τέτοιες ιστοσελίδες από απελάτες. Και τέλος, εξίσου όμως σημαντικό, είναι ότι θέλουμε να πετύχουμε ένα επίπεδο πρόληψης για εκείνους οι οποίοι υποτροπιάζουν και ιδίω για τα άτομα εκείνα τα οποία πηγαίνουν σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χώρα διαμονή του και προσπαθούν και εκεί να έρθουν σε επαφή με παιδιά για επαγγελματικού λόγου. Για παράδειγμα, όπω στην περίπτωση στην υπόθεση Φορνιρέ. Δηλαδή, άτομο το οποίο διώκεται ποινικά πηγαίνει σε μία άλλη χώρα και οι αρχές στη χώρα εκείνη δεν γνωρίζουν καθόλου ποιο είναι το ποινικό μητρό του ανθρώπου αυτού. Προσπαθούμε λοιπόν να βασιστούμε σε ένα σύστημα το οποίο στο σύστημα έκρηση, το οποίο αποφασίστηκε πρόσφατα για την ανταλλαγή στοιχείων ποινικού μητρώου από τη μία χώρα στην άλλη. Και κατά αυτόν τον τρόπο θέλουμε να εμποδίσουμε την περίπτωση εκείνη όπου σημαντικές πληροφορίες που θα έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την, ε, με την καταδίκη ενός ανθρώπου ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες και σε ένα άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή θα έχουν περάσει στο ποινικό μητρό του συγκεκριμένου ατόμου και θα έχουν ε, δοθεί στη συνέχεια σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η Προεδρία είναι σε θέση να σας πει περισσότερα πράγματα για το Πώ έχουν να κάνουν τα πράγματα με τις συζητήσει, πώς γίνεται η συζήτηση στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή στην ομάδα συμβουλίας για το ποινικό δίκαιο, η οποία συζήτηση είναι εξελίξη. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο τη Σουηδικής Προεδρίας, ο εκπρόσωπο θέλει να λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε Προβουλευτές... Είναι απόλυτα αληθές όπως το παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της ότι ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της τσεχικής προεδρίας είχε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για αυτή την ε, ρύθμιση. Η Σουηδική Προεδρία πήρε τη σκητάλη από την Προεδρία της Τσεχίας και τον Ιούλιο είχαμε μια πρώτη συνεδρίαση υπό την ηγεσία, υπό την πρωτοκαθεδρία από πλευράς της Σουηδίας ε, του Συμβουλίου. Μπορεί κανείς να πει ότι τα κράτη-μέλη αυτή την πρωτοβουλία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την χαιρέτησαν. Ήταν καλοδεχούμενοι. Ήταν θετικά διακείμενοι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών ενάντια αυτής της πρότασης. Πρόκειται εξάλλου και για ένα, μια προτεραιότητα η καταπολέμηση τέτοιου είδους αδικημάτων, τέτοιου είδους εγκλημάτων. Και πρέπει κανείς στην σημερινή απόφαση πλαίσιο να την προσαρμόσει και να την επικαιροποιήσει μια και αλλάζουν οι μέθοδοι εργασίας και η μεθοδολογία και ένα μεγάλο μέρος των αδικημάτων διαπράττεται μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Γίνονται περισσότερα ταξίδια από πλευρά των πολιτών μας, μεγαλύτερη κινητικότητα υπάρχει και έτσι η νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί αντίστοιχα. Από πλευρά των όσων ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εξάλλου σαφές εντωμεταξύ ότι Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για ένα ευρύτατο πεδίο δράσης, για ένα ευρύτατο θέμα και έχει μεγάλο φάσμα, ευρύτατο φάσμα αδικημάτων και έτσι θα πρέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων να θεσπιστεί. Αυτό χρειάζεται τον χρόνο του και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πλευρά, η χρονοβόρα πλευρά στην αποκαλέσω έτσι. Η Σουηδική Προεδρία τώρα τι θέλει. Η Σουηδική Προεδρία επιθυμεί να προαγάγει, να προωθήσει αυτές τις ε, διαβουλεύσεις και ή δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα χειροπιαστό τελικό αποτέλεσμα. Τώρα τούτων λεχθέντων ίσως θα μπορούσα να αναφέρω εν παρόδο ότι αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η ολοκληρωμένη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη είναι πολύ καλοδεχούμενη. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα ας ακούσουμε και από πλευράς του εισηγητή, της εισηγήτριας που την εκπροσωπεί ο Τζακολίνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως είπατε προηγουμένως αντικαθιστώ τη συνάδελφο Αντζελίλη η οποία λόγω πένθους χρειάστηκε να παραμείνει στην Ιταλία. τόσο το Συμβούλιο όσο και η Προεδρία έθεσαν σαφώς το ζήτημα αναθεώρησης του κειμένου του 2004. Πρόκειται για ένα σημαντικό αδίκημα, ένα από τα πιο βαριά και απεχθή αδικήματα τα οποία πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Ήδη τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και η, της, ε, ποινές που προβλέπει η συνάδελφος ε, τι ε, θεωρώ τις κατατάσσει σε πέντε επίπεδα. Ήδη μιλήσαμε για το grooming. θεωρείται ως αδίκημα η σεξουαλική εκμετάλλευση του ανήλικου ε, ε, και, στην, μέσα στην οικογένεια σε περίπτωση επίσης αποπλάνησης σε ε, αναμορφωτήριο απαγόρευση επίσης Ε, στην επαφή καταδικασμένων για δικήματα παιδοφιλίας ε, με ε, ανηλικούς και θα έλεγα ότι σε αυτά που ήδη αναφέρει η συγγήτρια πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Θα πρέπει να προσθέσουμε την ψυχολογική βοήθεια από τον, ψυχολόγο να μπορέσουμε να έχουμε και την δυνατότητα της προσφυγής σε παιδοψυχίατρο. Χρειάζεται λοιπόν υποστήριξη επίσης και από νομικής πλευράς Και τελευταίο προτείνουμε έναν ευπρεπή τρόπο ζωής στην οικογένεια. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται κατάρτιση σε επίπεδο οικογένειας και να ενισχύονται οι διάφοροι οργανισμοί οικογενειακής υποστήριξης ούτως ώστε να προλαβαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα αποπλάνησης των ανηλίκων. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε καθυστερήσει όμω σε σχέση με το αρχικό μα χρονοδιάγραμμα. Σα παρακαλώ λοιπόν πολύ να είστε σύντομοι στι παρεμβάσει σα. Η κυρία Σίπελ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα έλεγα αυτό το πρόβλημα το ότι το ξαναβλέπουμε και το ξανασυζητάμε είναι αρκετά αρνητικό. Χαίρομαι όμως ότι στην έκθεση γίνεται η προσπάθεια οι τεχνολογίες επικοινωνίας να χρησιμοποιηθούν και να γίνει η προσπάθεια να υπάρξουν ρυθμίσεις ώστε η διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας να αναχαιτιστεί, να περιοριστεί. Ωστόσο πιστεύω ότι από πλευράς ε, της αναχέτησης αυτής ε, ε, δεν θα έχουμε τελεσίδικα αποτελέσματα. Είναι μεγάλη η δυνατότητα να παρακάμπτουν τέτοιου είδους φραγμούς ή περιορισμούς. Είναι τόσο θα έλεγε κανείς απλό κάτι τέτοιο ώστε δεν μπορεί κανείς να περιμένει αηφόρο αποτέλεσμα από κάτι τέτοιο. Για τα παιδιά που αφορώνται εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε πιστεύω ότι οι αντίστοιχε σελίδε πορνογραφικού υλικού για παιδιά πρέπει να αφαιρεθούν από το διαδίκτυο. Μπορεί αυτό να γίνεται μια και τα κράτη θα πρέπει να υποχρεούνται να κάνουν κάτι και να μην ανέχονται αυτά. Όμως από υπερπόντια σημεία υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, τέτοιου είδους ε, δικτύων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι από υπερπόντια τέτοια σημεία δεν θα υπάρχει διοχέτευση τέτοιου υλικού. Μόνο η φραγή του υλικού δεν θα είναι δυνατόν να αποφέρει αηφόρα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης ε, και την ε, Προεδρία, τη Σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που μπορώ να προσθέσω τη φωνή μου εγώ εδώ και να πω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό τομέα απέναντί μας. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέτοιες καλές θετικές προτάσεις που αφορούν όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής. Όμως θα ήθελα ακριβώς σε αυτό το ένα σημείο να τονίσω κάτι. Φραγή διαδικτύου, όπου έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κίνδυνος εδώ, οι καλές προθέσεις μας, οι καλές προτάσεις με μια, ας το πω έτσι, βιαστική δράση να υποβαθμιστούν, να διακυβευθούν. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω που θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά από πολλά άλλα, τα οποία λένε να μην γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, να μην τύχει συνέχεια. Αφενό είναι το ότι εμεί ω Ευρωβουλή επανειλημμένα έχουμε πει ότι ουσιαστικά η διεθνή συνεργασία για την πραγματική δίωξη και για την απάλληψη, κατάργηση αυτών των σελίδων στο διαδίκτυο αυτού του πορνογραφικού περιεχομένου πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας και πρέπει πολύ πιο έντονα να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Αν δει κανείς το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για παράδειγμα, η επιβολή, νομική επιβολή της απάλληψης αυτού αυτών των θεμάτων έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι σε σχέση με τα παιδικά δικαιώματα ή τα θέματα αυτά, συναφή θέματα. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν περισσότερο σε αυτόν τον τομέα, να κάνουμε κάτι παραπάνω επιτέλους, ώστε τα κράτη με σαφή τρόπο να υποχρεωθούν να σβήνουν, να απαλήφουν αυτές τις σελίδες. Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι οι φραγές θα είναι αποτελεσματικές. Σημαντικό είναι να ξέρει κανείς ότι το μεγάλο μέρος, μεγαλύτερο μέρος ε, αυτού του υλικού, του παιδικού πορνογραφικού υλικού δεν είναι στη διάθεση των σερφερ εκεί σε χώρες όπου δεν υπάρχει νομική εποπτεία, αλλά βρίσκεται εκεί όπου έχει ισχυρούς εμπορικούς εταίρους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί όπου στους άλλους τομείς λειτουργούν τα πράγματα, εδώ όμως σε αυτόν τον τομέα που θα έπρεπε να λειτουργούν για την παιδική πορνογραφία, πολύ λίγα γίνονται για εναλλακτικέ λύσεις και για την αναζήτηση αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων και την ε, αποσαφήνισή τους. Και έχω την εντύπωση ότι ουσιαστικά στην αξιολόγηση και αποτίμηση αυτών των μέτρων όσον αφορά την, ε, ε, το σκόπιμο φραγών στο διαδίκτυο, όσον αφορά το αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή όχι, αν υπάρχουν κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις που είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και στον τομέα της σκοπιμότητας δηλαδή βλέπουμε ότι οι φραγές στο διαδίκτυο δεν είναι πολύ αποτελεσματικές και δεν φέρνουν και σε σχέση με τα πραγματικά τεκμήρια ή αποδείξεις χωλένουν τα πράγματα και υπάρχει απουσία τεκμηρίων ή αποδεικτικών στοιχείων και έτσι είναι απόλυτα ασαφές σε ποια βάση βασίζονται τέτοιες ε, δράσεις και στην ε, αποτίμηση επιπτώσεων δεν υπάρχει κάποια αξιολόγηση και έχω την εντύπωση ότι εδώ θα έπρεπε να διερωτηθούμε και να προβληματιστούμε. Όταν έχουμε τόσες καλές προτάσεις και προθέσεις φαίνεται εδώ το ζήτημα να είναι περισσότερο αν στο θέμα της επιβολής σε νομικό πλαίσιο για το διαδίκτυο μπορεί να επιτευχθεί κάτι για την απάλληψη τέτοιων σελίδων, τη διαγραφή τους ή αν πρόκειται για συμβολική σημασία μέτρα τα οποία έχουν μάλλον βιαστικό χαρακτήρα και δεν είναι τα πιο σκόπιμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς τώρα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όπως πολλοί άλλοι προλαλήσαντες ανέφεραν, Πρόκειται εδώ για τα χειρότερα δικήματα εγκληματικής μορφής και πρέπει αυτή την τρομερή κατάσταση, αυτό το αποτροπιαστικό πράγμα να το καταπολεμήσουμε από κοινού. Θέλω να πω καταρχήν ότι θεωρώ θετική αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει κάτι να κάνουμε, είναι σαφέστατο αυτό. Έχουμε διαβάσει εξάλλου και στο έγγραφο ότι εκείνο που θέλουμε είναι να κλείσουν αυτές οι σελίδες του διαδικτύου να μην είναι προσπελάσιμες όμως πιστεύω ότι κατά πρώτο λόγο πρέπει να λάβουμε υπόψη τα παιδιά. Τα παιδιά να θέσουμε στο επίκεντρο και παγκόσμια. Πρώτα να λάβουμε υπόψη το συμφέρον των παιδιών. Να βρούμε τα παιδιά τα οποία εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Μπορεί να κλείσει κανείς χιλιάδες, μυριάδες σελίδες στο διαδίκτυο. Όμως ταυτόχρονα Μυριάδες παιδιά υφίστανται τα πάνδυνα από τέτοιου είδους μηνύματα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν αυτά τα παιδιά, να ανοιχνεύσουμε αυτά τα παιδιά, να τα ταυτοποιήσουμε. Έχω λοιπόν αμφιβολίες σχετικά. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς το Συμβούλιο. Όταν ακούσαμε τις ε, επεξηγήσεις του Συμβουλίου και τις τοποθετήσεις αναφέρθηκε ότι χαιρετίζεται λέει και είναι καλαδεχούμενη αυτή η πρόταση ότι με θετικό πνεύμα την αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη κάπως όμως ε, έγινε κατανοητό, αφέθηκε να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Θα ήθελα να ξέρω κάτι παραπάνω για αυτά. Είναι λοιπόν πραγματικά τόσο καλή αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πείτε μας πώς διεξάγεται η συζήτηση στο Συμβούλιο γύρω από αυτήν και τώρα και την τελευταία φορά στο Στρασβούργο είχα και μία ερώτηση προς την Σεσίλια Μάρστροεμ την οποία είχα διατυπώσει. <clears throat> Η Σουηδική Προεδρία πώς βλέπει αυτά τα θέματα της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και του σεξοτουρισμού. Τα βλέπει ως μια προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας. Θα έπρεπε να γίνει λοιπόν μια ε, ακρόαση για την Ευρώπη των παιδιών στις 20 Νοεμβρίου. L'Europe des enfants, η Ευρώπη των παιδιών. Και αυτό το θέμα ακριβώς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών ήθελαν να το εξετάσουν με το σεξοτουρισμό, σεξουαλικό τουρισμό. Άκουσα όμως εντωμεταξύ δεν συμβαίνει λέει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ερώτηση προς το Συμβούλιο αυτό το σημαντικό θέμα. Δεν θα εγγραφεί λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Romeva. Κύριος No. Δεν θέλετε να παρέμβετε. Mrs. Romero. Κυρία Ρομέρο, παρακαλώ. Ρομέρο. Ρομέρο. Then... Όχι. Εντάξει, κύριος Μπουσούτη λοιπόν, παρακαλώ. Eh, eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω επίση να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι παρεμβάσει του. Και θέλω επίση να ευχαριστήσω για την, για την παρέμβαση του κυρίου Γιακολίνο για αυτό το θέμα. Θα έλεγα όλοι οι γονεί έχουν τον ίδιο, του ίδιου φόβου. Ο μεγαλύτερο φόβο του είναι τι θα γίνει με τα παιδιά του που εκτίθενται στο διαδίκτυο σε τέτοια μηνύματα και ποιοι κίνδυνοι αναμένουν τα παιδιά στο διαδίκτυο Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι πρέπει να λάβουμε κάθε μέτρο, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και μάλιστα με κατεπήγοντα τρόπο, κατεπηγόντος, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να προσφέρουμε στα παιδιά μας την προστασία εκείνη παντού και πάντα όπου, την χρειάζονται. Ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους καταστάσεις όπου διακυβεύεται η σεξουαλική τους εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευσή τους ως αντικειμένου για πορνογραφικούς σκοπούς. Μία ερώτηση θα είχα. Ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων μας στο επίπεδο των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αν δεν κάνω λάθος αυτό αφορά το ποινικό ε, δίκαιο και τον εναρμονισμό των δράσεών μας όσον αφορά το ποινικό δίκαιο και την ποινική ε, νομοθεσία και την ποινική δικονομία για αυτά τα θέματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ή εκπρόσωπος θα μπορούσε να μας πει ποια είναι τα όρια των δικών μας αρμοδιοτήτων σε τέτοια θέματα. Και να δούμε επίσης Μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο εμείς με βάση τις αρμοδιότητες μας ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Διατυπώνω αυτή την ερώτηση διότι γνωρίζω ότι κάποιες ε, αποφάσεις ε, από πλευρά νομολογίας του ΔΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν ληφθεί από πλευράς ε, του που θέτουν περιοριστικά όρια με αυστηρό πνεύμα μέχρι πού μπορεί κανείς να φτάσει σαν εμάς σε αυτό το επίπεδο. Σε ευχαριστώ. Ματιέ παρακαλώ. Ματιέ. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις για αυτό το τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Το πρώτο αφορά στην πρόληψη. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε περισσότερη πρόληψη στο θέμα. Δυστυχώς όταν γνωρίζουμε ότι τα θύματα πολλές φορές ε, γίνονται θύτες όταν μεγαλώνουν. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει πρόληψη έναντι αυτών των παιδιών και για τον σεξουαλικό τουρισμό. Θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν έχει στοιχεία για αυτού του τύπου τον ε, τουρισμό, εκτός φυσικά ευρωπαϊκών ε, συνόρων, γιατί εγώ είχα πάει στην Καμπότζη κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και είχα εντυπωσιαστεί ο σεξουαλικός ε, τουρισμός από την Ευρώπη ήταν πάρα πολύ σημαντικός στην ε, Καμπότζη και ξεπλάγει όταν τα μέλη της Ευρω... Ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων μου λέγανε ότι οι Ασιάτες είναι οι μεγάλοι καταναλωτές παιδιών και κυκλοφόρησα τέλος πάντων σε διάφορα ύποπτα ε, μέρη για να δω τι γίνεται. Είδα με τα μάτια μου τι συμβαίνει και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μου το επικύρωσαν. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι έχει γίνει από αυτού. Κύριε Έλστ. Η ε, κυρία Έλστ, ευχαριστώ πολύ. Στα τσεχογερμανικά σύνορα με απασχόλησε αυτό το θέμα επί αρκετά χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ καλό να κάνουμε κάτι για την προστασία των θυμάτων, να το κατοχυρώσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και το χαιρετίζω. Εκείνο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει ακόμα να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί είναι θέματα της πρόληψης και της δουλειάς σε σχέση με τους ε, δράστες δουλειά όσον αφορά τους ίδιους τους δράστες, ώστε περαιτέρω τέτοια αδικήματα, τέτοια εγκλήματα να αποφευθούν, να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε με επίκεντρο αυτό το θέμα για να ανταποκριθούμε με το σωστότερο τρόπο σε αυτό το καθήκον. Έχω μια αμηχανία, δύσκολη ας το πω έτσι τοποθέτηση αμφίροπη θέση όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Στην Γερμανία είχαμε επί πολλά χρόνια αυτή τη συζήτηση. Ποινικό δίκαιο. Να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει από αυτό. Όχι να οξύνουμε, να κάνουμε αυστηρότερες τις ποινές, αλλά να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο. Δηλαδή, αυτό έχει επιπτώσει στα παιδιά. Δηλαδή, όλο και χειρότερα εγκλήματα και πιο ε, αποτροπιαστικά εγκλήματα γίνονται. Και γι' αυτό το αίτημα να είναι αυστηρότερες πάντα οι ποινές πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Είναι αυτή η σωστότερη πορεία. Μπορούμε να κατοχυρώσουμε έτσι την σωστότερη δράση. Το τρίτο σημείο που είναι σημαντικό είναι το θέμα της ε, αστυνομικής συνεργασίας. Και εδώ στην αστυνομική συνεργασία υπάρχουν μεγάλε ελλείψεις. Το είδα σε αυτή την περιφέρεια εκεί που προανέφερα. Η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί για την καταδίωξη τέτοιων εγκλημάτων ει βάρο των παιδιών. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό που πρέπει πολύ περισσότερο να υπογραμμιστεί και να ενταθεί. Και τελευταίο, το προανέφεραν οι συνάδελφοι, η φραγή στο διαδίκτυο δεν δίνει αποτελέσματα. Είχαμε πολλά χρόνια συζήτηση με πινακίδε και με σήματα ε, για φραγές δεν είναι η σωστή πορεία αυτή. Πρέπει και πάλι να ξανασκεφτούμε πώς θα σβήνουμε σελίδες, θα τις απαλήφουμε ώστε αυτό το θέμα πιο καταλεπτός, πιο εξειδικευμένα να αντιμετωπιστεί. Να μην κάνουμε κάτι το βιαστικό το οποίο δεν θα είναι αποτελεσματικό. Να πάρουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεγιόν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνεχίζοντας εγώ σε αυτά τα οποία προανέφερε η κυρία Έρνστ, θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο είναι κάτι γενικότερο. Πρόκειται και πάλι για μια πρόταση εδώ που ένα τμήμα, ένα μέρος του ποινικού δικαίου εναρμονίζεται. Για τους καλύτερους λόγους βέβαια. Γιατί είμαστε φυσικά υπέρ η κακοποίηση των παιδιών να καταπολεμάται πάντα και να καταπολεμηθεί σε όλα τα επίπεδα και με μεγαλύτερη εντονότερη συνεργασία. Αυτό όμως που απουσιάζει σε αυτή την impact assessment, την αποτίμηση επιπτώσεων, είναι το πώς έχουν τα πράγματα για τον εναρμονισμό του ποινικού δικαίου και της ποινική δικονομίας. Λείπει εδώ η θέση, το στοιχείο διασύνδεσης αυτού του θέματος και αυτού που επιθυμεί ο Επίτροπος Μπαγό. Θέλουμε πραγματικά έναν εναρμονισμό του ποινικού δικαίου. Ο κύριος Μπαρό λέει όχι γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν οριμάσει επαρκώς και δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Κάτι έχει υπόψη τη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι λοιπόν ο τελικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής εδώ. Είναι επικίνδυνο πάντα να εναρμονίζεται ένα τμήμα έστω του ποινικού δικαίου αλλά πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εναρμονίζονται και να μην ρυθμίζονται. Η κακοποίηση των παιδιών ναι να εναρμονιστεί διότι πολλά από αυτά τα εγκλήματα, τα αδικήματα συναρτώνται και συνδέονται το ένα με το άλλο. Αν θέλουμε ένα ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο τότε προστίθεται σε αυτό το θέμα ως ζητούμενο τι πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ρυθμίσουμε και εσύ τι στο επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό η impact assessment δεν επαρκεί για αυτή την πρόταση η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Δεν επαρκεί αυτό Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια ποια κατεύθυνση στοχεύει να ακολουθήσει το ποινικό δίκαιο ή, ε, το εγχείρημα αυτό και τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι θα γίνει σε επίπεδο κρατών μελών και πώς συσχετίζεται αυτή η πρόταση εδώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον γενικό εναρμονισμό του ποινικού δικαίου. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει κοινή νομοθεσία για κυρίαρχα κράτη. Πάντως, σαφώ θα ήμουν υπέρ τη απαγόρευσης κατανάλωση τη παιδική πορνογραφία με μηδενική ε, ανοχή. Θα μπορούσα λοιπόν απόλυτα να συμφωνήσω με την απαγόρευση στο σελίδων με το φραγμό των ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας. Αυτό θα με έβρισκε απόλυτα σύμφωνη. Θα ήμουν σύμφωνη επίσης με την απαγόρευση κατοχής υλικού παιδοπορνογραφικού και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάποιοι συνάδελφοι έχουν, έχουν προβλήματα με την νομική βάση. Ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί να σκέφτονται κάπως διαφορετικά. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής πίσω από κάθε υλικό παιδο πορνογραφικό κρύβεται ουσιαστικά ένα έγκλημα. Ένα πολύ σοβαρό έγκλημα, από τα πιο σοβαρά έγκληματα που θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ κανείς. Δεν πρόκειται για απλά σύμβολα. Ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα πραγματικά παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, που υπέφεραν προκειμένου να δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα, προκειμένου να δημοσιευθεί μια φωτογραφία τους και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η απαγόρευση που εμείς προτείνουμε. Είναι απόλυτο νόμιμο, απόλυτα νόμιμο το να καταφέρουμε να διώξουμε την, τη ζήτηση προκειμένου να καταφέρει να μειωθεί και η προσφορά. Είναι σημαντικό να ποινικοποιούνται και να διώκονται όχι μόνο αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το υλικό αυτό, αλλά και αυτοί που καταναλώνουν το παιδοπορτογραφικό υλικό. Ότι και τα άτομα αυτά, οι καταναλωτέ δηλαδή, είναι αναπόσπαστα στοιχεία της όλης αλυσίδας χωρίς ε, τη δική τους ουσιαστικά ζήτηση για αυτό το προϊόν δεν θα υπήρχε και η προσφορά αυτού του προϊόντος. Χωρίς τη δική τους συμμετοχή στην αλυσίδα αυτή δεν θα υπήρχε και η δημιουργία πορνογραφικών, παιδοπορνογραφικών ιστοσελίδων. Ας μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε εικόνα που βλέπετε στο ίντερνετ κρύβεται ένα παιδί το οποίο υποφέρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου κάθε φορά, το οποίο, κάθε φορά που μιλάμε για παιδική πορνογραφία και λυπάμαι που ο συνάδελφο από τη Γερμανία γελάει, γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσο φιλελεύθεροι και να είμαστε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε ε, το να υποφέρουν τα παιδιά. σα. ευχαριστώ πολύ. Άλλε παρατηρήσει από τον κύριο Άλμπρεκτ. Ίσως. Με παρανοήσατε. Ίσως το κατέστησα σαφές ότι μου είναι εξίσου σημαντικό εμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν να υποβάλουν αυτή την πρόταση κατά του πορνογραφικού υλικού που πρέπει να καταπολεμηθεί. Δεν είναι καθόλου πρόθεσή μου εδώ να συνεργαστώ ώστε να υπάρχει χαλαρότερη θέση και μικρότερες προσπάθειες κατά της παιδικής πορνογραφίας. Το αντίθετο, εκείνο όμως που θέλω εγώ είναι αυτή η πρόταση σε αυτό το σημείο να δούμε ότι είναι κάτι το βιαστικό με την, το κλείσιμο σελίδων στο διαδίκτυο. Όχι ότι εγώ δεν θέλω να εξαφανιστούν αυτές οι σελίδες από το διαδίκτυο, διότι και εγώ το θεωρώ εξίσου σημαντικό όπως και εσείς να μην παράγονται τέτοιες σελίδες και να μην διαχέονται, να μην διαδίδονται στο διαδίκτυο με σελίδες εκεί αλλά θέλω να δούμε ποια προσέγγιση θα υιοθετήσουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα σβήσουμε αυτέ τι σελίδε ή θα θέσουμε φραγέ μόνο. Πράγμα το οποίο είναι επιφανειακή, αν θέλετε, επιφανειακό περιορισμό και όχι αποτελεσματικό ε, τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με εκείνου που ανταλλάσσουν τι σελίδε αυτέ. Αφορά, για παράδειγμα, κάτι που μπορεί κάποια σελίδα να κλείσει. Ε, που ίσως ε, σε σχέση με την, ε, τα περαιτέρω μέτρα από την ε, φραγή είναι ένα είδος λογοκρισίας πάντα θα πρέπει να εξετάζεται αν, είναι, ενδεικνύεται ένα τέτοιο μέσο και αν είναι πραγματικά σκόπιμο να αναλαμβάνετε τέτοια πρωτοβουλία. Δεν έχει καμιά σχέση με το, θέλουμε, με το ότι θέλουμε όλοι να προστατέψουμε τα δικαιώματα των παιδιών με τη δράση μας, που πρέπει να γίνει σίγουρα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Στρεφόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαρινάρο, παρακαλώ η κυρία Μαρινάρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι Σίγουρα θα μπορούσα να δώσω καλές απαντήσεις σε όλες αυτές τις πολύ καλές ερωτήσεις που ακούστηκαν και στα σημαντικά ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι ευρωβουλευτές. Εναλλακτικές λύσεις όντως εξετάσαμε, ναι. Χρησιμοποίησαμε πυραγνωμοσύνη, τεχνογνωσία όταν καταρτίζαμε την πρόταση αυτή. Χρησιμοποίησαμε ιδιαίτερα την εμπειρία της Ευρωπόλ η οποία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο τομέα της ε, παιδικής πορνογραφίας και γενικότερα στα πλαίσια της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών. Και η πυρογνωμοσύνη βέβαια υπάρχει και σε μονομένα κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο όπου ε, η ΣΥΟΠ είναι μια υπηρεσία ιδιαίτερα δραστήρια στην, στο Ηνωμένο Ανάλογη υπηρεσία υπάρχει και στην Ιταλία, ιδιαίτερα δραστήρια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπήρχε εδώ πέρα μία μόνο δράση που θα αποτελούσε την μαγική λύση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τεχνολογία είναι παρούσα, είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να καταπολεμήσει κανείς τέτοιες καταστάσεις, αλλά το να κλείσουμε απλώς ένα διαδίκτυο, ένα, μια ιστοσελίδα, ένα ιστότοπο, είναι φύση αδύνατο, γιατί ο ιστότοπος αυτός ενδεχομένω να μην βρίσκεται καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να επεκτείνουμε τη δικαιοδοσία, την ποινική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός και σε τρίτες χώρες, προκειμένου να είμαστε σε θέση να κλείνουμε ιστο, ιστοτόπους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Βέβαια γνωρίζουμε ότι στην πράξη κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δράση την οποία η δράση η την οποία υιοθετούμε ενδεχομένω να μην είναι απόλυτα αποφασιστική και να μην αποτελεί μια μαγική λύση, αλλά σίγουρα μπορεί να συμβάλλει. Ενδεχομένω δηλαδή να μειώσει τα κέρδη των ανθρώπων αυτών που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ιστοσελίδες, των ιδιοκτητών των ιστοσελίδων αυτών. Προσπαθούμε λοιπόν να εξετάσουμε μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών δράσεων. Για παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει ένα financial collision, έτσι το ονομάζουμε, ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα μία σύμπραξη που έχει να κάνει με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με συνεργασία πιστοτικών φορέων, τραπεζών και άλλων οργανισμών πληρωμής όπως το PayPal και η βασική εδώ ιδέα είναι να καταφέρουμε να ανοιχνεύσουμε την πορεία που ακολουθούν τα χρήματα, μία πληρωμή δηλαδή για υλικά παιδικής πορνογραφίας και να καταφέρουμε να δώσουμε τέλος στη σύμβαση αυτή χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία έχει στη θέση της μία τράπεζα. Σας το λέω αυτό για να σας πω ότι η νομοθεσία δεν αποτελεί πανάκια, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό τμήμα μιας πιο πολύπλοκης δράσης. Δεύτερον, ταυτοποίηση των παιδιών. Σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ορισμένε μη κυβερνητικέ οργανώσει θεωρούν ότι η παιδική πορνογραφία δεν θα πρέπει να ονομάζεται child pornography αλλά sexual abuse images, δηλαδή εικόνε παιδική εκμετάλλευση, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και όντω πίσω από κάθε εικόνα παιδικής πορνογραφίας κρύβεται μία περίπτωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Και σίγουρα τα παιδιά αυτά που πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα για μας. Γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε και, με, και στα πλαίσια αυτής της χρηματοοικονομικής συμφωνίας σύμπραξης του Financial Coalition στο οποίο αναφέρθηκα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι συντάξαμε την πρόταση αυτή ε, όντας σε απόλυτη διαβούλευση με τη νομική μας υπηρεσία, έχουμε ελέγξει κάθε νομική διάταξη της πρότασης αυτής και η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η κάθε διάταξη που χρησιμοποιούμε συνάδει με την ε, νομική βάση, γιατί κάθε διάταξη ουσιαστικά καλύπτει τον ε, πρωταρχικό στόχο που είναι η προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Όσον αφορά τα μέσα στα οποία αναφερθήκατε, δεν έχω να σας δώσω συγκεκριμένα δεδομένα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο εντελώς ε, υπόγειο, κρυφό, δεν ε, υπάρχει δυνατότητα της ε, καταδίωξης, ε, της ποινική διερεύνησης όλων αυτών των περιπτώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες δεν τιμωρούνται τελικά στα περισσότερα κρατημέλα, ακριβώ επειδή δεν εντοπίζονται. Ευχαριστούμε πολύ, Σουηδική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντικό και μετά από τα όσα είπε ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από αυτό που έθιξαν πολλοί προλαλήσαντες, δηλαδή το θέμα των φραγών στο διαδίκτυο, των σελίδων στο διαδίκτυο. Φυσικά μπορεί να διαρωτηθεί κανείς πόσο αποτελεσματικό είναι ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά να δούμε και το ότι μπορεί να το δει κανεί από μια άλλη προσέγγιση, από μια άλλη γωνία και μέσω του συστήματο πληρωμή ή συνδρομών, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο να το προσεγγίσει κανεί για να είναι πιο αποτελεσματικό. Διατυπώθηκε η παράκληση να ακούσετε κάτι παραπάνω τι λένε τα κράτη-μέλη για αυτή την πρόταση από πλευρά του ή τι είπαν. Πώς αξιολογούν τα πράγματα δηλαδή τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, προσέξτε, πρόκειται για περίπλοκα, σύνθετα θέματα και δεν είναι απλό όλα όσα προτείνονται σε αυτή την απόφαση πλαίσιο από τα κράτη-μέλη να γίνουν δεκτά τα πάντα χωρίς καμία επιφύλαξη ή δεν θέλω να πω ότι όλοι έχουν την ίδια προσέγγιση και την ίδια άποψη απόλυτα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τώρα είναι υπερβολικά πρόημη πρόωρη η στιγμή χρονικά για να, να πει κανείς ή να ταξινομήσει ποιε είναι οι θέσεις του Συμβουλίου ή πώς επιμερίζονται οι τοποθετήσεις. Ο πρώτος γύρος διαβουλεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν και θα επανέλθουμε στο μέλλον σίγουρα για να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θεωρούν από πλευρά τους ότι μπορεί να υιοθετήσουν μια θετικότερη προσέγγιση. Με άλλα λόγια, σε σχέση με την επανεξέταση των κυρώσεων, να υπάρχει καλύτερη, μεγαλύτερη αναλογικότητα, να είναι πιο αποτελεσματικές οι ποινές και οι κυρώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί από τις μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις. Τα κράτη-μέλη εκείνο που γενικά κάνουν είναι εκφράζουν την άποψη ότι πρέπει να επανέλθουμε και πάλι να ξαναδούμε τις προτάσεις του 2002. Σας ευχαριστώ. Ναι, και κάτι άλλο. Ξέχασα κάτι. Υπάρχει και ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσω και να επανέλθω στη συνέχεια, γιατί τώρα δεν μπορώ να δώσω ακόμα κάποιο σημείο. Γιατί αυτό το σημείο στην διάσκεψη του Νοεμβρίου, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει εγγραφεί εκεί στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Είχαμε λοιπόν μια εκτενή και ζωντανή συζήτηση και για κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις επανερχόμαστε στον κύριο Τζακολίνο παρακαλώ. Mi pare che il ε, dibattito abbia consentito di affermare intanto una ε, ε, ε, μου φαίνεται ότι από τη συζήτηση προκύπτει μία βεβαιότητα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή και πνευματική διάβια. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που μπορούμε να συμμεριστούμε. Σίγουρα λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε με όλες τις συνεισφορές ε, των συναδέλφων εδώ στην αίθουσα. Πρόεδρος, νομίζω ολοκληρώνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, σίγουρα, και νομίζω ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που είναι προτεραιότητα, μία από τις προτεραιότητες στην ευαισθησία όλων των μελών στην Ευρωβουλή και αυτό έχει επίπτωση σίγουρα στα ίδια τα θεμέλια αυτό το θέμα. Στην ποινική νομοθεσία των, των κρατών μελών μας. Σίγουρα. Αυτό ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και έχοντας μια τόσο ζωντανή συζήτηση που ολοκληρώσαμε, φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποιο πρόσθετο στοιχείο του, από τον κύριο Ντεγιόγκ, παρακαλώ. Θέλετε να παρέμβετε, έχετε τον λόγο. Ναι, λυπούμε, συγχωρήστε με πρόεδρε που ζητώ να, να παρέμβω πάλι. Είχα μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν απαντήθηκε. Ήταν και ένα δύσκολο ερώτημα για τον εναρμονισμό σε γενικά πλαίσια του ποινικού δικαίου. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να σημειώσει την ερώτηση και να την διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε υστερότερα να μας υποβληθεί γραπτός απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς έχει ο εναρμονισμός του ποινικού δικαίου γενικά σε γενικότερα πλαίσια και πώς σκοπεύουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσουν αυτόν τον εναρμονισμό. Θα μας διευκολύνει το έργο μας στο μέλλον αν μας δοθεί απάντηση σε αυτό. Κυρία Μαρινάρο, παρακαλώ. Δυστυχώς δεν είμαι αρμόδια για να δώσω απάντηση σε μια τόσο γενική ερώτηση. Σε γενικέ γραμμέ, στόχο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προφανώς είναι να προωθήσει την προσέγγιση του ποινικού δικαίου και των ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο γενικός αυτό στόχο αντανακλάται και στην πρόταση αυτή που συζητάμε. Βέβαια, δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση σε μια τόσο γενική ερώτηση. Λυπάμαι. Σα ευχαριστούμε. Νομίζω ολοκληρώσαμε με αυτό το συγκεκριμένο σημείο στην ημερησία διάταξη. Όλοι γνωρίζουμε ότι καθυστερούμε κάπως. Έχουμε κάποια καθυστέρηση. Πιέζει ο χρόνος. Είναι 5 και 20 και θα έλεγα ότι έχουμε τρία σημεία που πρέπει ακόμα να καλύψουμε Λοιπόν, είμαστε αναγκασμένοι να επιταχύνουμε κάπως τις διαργασίες. Το επόμενο σημείο είναι το σημείο 13 στην ημερησία διάταξη. Η πρόληψη και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων. Έχουμε εδώ σε αυτό το σημείο μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων μετά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα, πρέπει να καλωσορίσουμε ανάμεσά μας τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών ΦΑΜ που δέχτηκαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Η Σουηδική Προεδρία επίσης την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων τη θεωρεί ως μια κυρίαρχη πρωταρχική προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας. Συνεχίζονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο για μια απόφαση πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, η απόφαση πλαίσιο που ε, υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με απόρριψη λόγω έλλειψης χρόνου στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών η συζήτηση αυτού του ευαίσθητου θέματος αναβλήθηκε για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Δρατώμεθα λοιπόν της ευκαιρίας να σας υπενθυμίσουμε ότι ζήτησε το Συμβούλιο από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει επ' αυτού μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2009. Αν η συνθήκη της Λισαβόνας αρχίσει να ισχύει, εγκριθεί και αρχίσει να ισχύει, αυτή η πρόταση θα αλλάξει νομική βάση και η Ευρωβουλή θα εμπλέκεται στη διαδικασία συναπόφασης ως συνομοθέτης. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, σας προτείνω να ξεκινήσουμε λοιπόν, δίνοντας τον λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Χέντ, και στη συνέχεια θα έχουμε την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την εκπρόσωπο της Σουηδικής Προεδρίας. Κυρία Χέντε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Προσέξτε, προσέρχομαι εδώ, έρχομαι σε ένα περαιτέρω σημαντικότατο θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η εμπορία ανθρώπων ανήκει στα πιο αποτροπιαστικά εγκλήματα Απαγορεύτηκε επίσημα στο παρελθόν αυτό το έγκλημα. Εδώ και 200 χρόνια η σκλαβιά, η δουλεία. Όμως 200 χρόνια μετά Μιλιάδες άνθρωποι πλήττονται από αυτή το, αυτό το είδος δουλείας, δηλαδή από την εμπορία ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα θεσμικά όργανα έχουν τεράστια ευθύνη αυτή την σύγχρονη μορφή δουλείας να την τροχοπεδίσουν, να αναχαιτήσουν, να την περιορίσουν. Έχουμε μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που είναι καλή αφετηρία, είναι πολύ καλύτερη από την παλαιά απόφαση πλαίσιο και για την συμφωνία επ' αυτού μπορούμε κάτι να πετύχουμε αν συμφωνήσουμε αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο από την δίωξη σε ποινικά πλαίσια θα έλπιζα ότι θα υπήρχαν πολλά περισσότερα προληπτικής μορφής μέτρα και πώς από κοινού αυτό το, αυτό το διασυνοριακό πρόβλημα, αυτή τη μάστιγα μπορούμε να την καταπολεμήσουμε. Σεξουαλική δουλεία, καταναγκαστική εργασία, η καταναγκαστική υιοθεσία σαν αποτέλεσμα αυτής της εκμετάλλευσης. Στρέφομαι λοιπόν σε ένα πρώτο ερώτημα σε σχέση με αυτό ο τίτλος αυτής της ε, απόφασης είναι «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων». Αυτό είναι ο ακριβής τίτλος της απόφασης ε, πλαισίου. Πρόκειται σε πρώτη γραμμή για την ποινική δίωξη όμως. Δεν πρόκειται τόσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Ή μήπω θα έπρεπε να λέγεται ποινικά μέτρα για την προστασία θυμάτων και τίποτα παραπέρα. Διότι κατά τα άλλα με ένα τέτοιο τίτλο θα μπορούσε να είναι παραπλανητικός και να απογοητεύσει κάποιους, να δημιουργηθεί ένα είδος απογοήτευσης γιατί δεν είμαστε ευρύτεροι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεύτερον, κάποτε στο μέλλον ερώτηση θα κάνουμε λόγο και για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων. Διότι αυτό απαιτεί σε μεγάλο βαθμό διασυνοριακή συνεργασία. Έχω φυσικά πολλές απόψεις, πολλές προτάσεις. Δεν θέλω όμως τώρα να εξαντλήσω και να παρουσιάσω τα πάντα. Ένα ερώτημα να θέσω. Αν δει κανεί το άρθρο 3 όσον αφορά ποινέ, κυρώσει και επιβαρυντικέ περιστάσει, τότε παρατηρεί κανεί εγκλήματα ει βάρο παιδιών υπό το 3-2 μέγιστη ποινή 10 έτη ε, καταρχήν θα έπρεπε οι ποινές, ε, τα αδικήματα έναντι παιδιών στο 3-3 να εντάσσονται. Στο 3-3, διότι εκεί απαιτούνται ελάχιστες ποινές 12 διάρκειας, 12 ετών. Κατά τα άλλα, οι ποινές υπό το 3,3 εις βάρος των παιδιών θα πρέπει να κατοχυρωθούν και να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι υπό αυτό τον τίτλο θα εντάσσονται οι ποινές. Πρόκειται για παιδιά που όλη τους τη ζωή τα διώκει αυτό το τραύμα αυτής της εμπειρίας, της τραυματικής εμπειρίας. Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή, να ανακούσουμε και από το Συμβούλιο τι γίνεται σε σχέση με την ε, παρακολούθηση αυτών των θεμάτων. Ποια επιμόρφωση, ποια εκπαίδευση, παιδεία θα δοθεί σε αυτά τα παιδιά στα παιδιά για τα θέματα αυτά της εμπορίας ε, ανθρώπων και παιδιών. Πώς θα υπάρξει η αντίστοιχη παιδεία και εκπαίδευση. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί μέσα στο πλαίσιο της λήψης απόφασης. Πώς αντιμετωπίζει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα. Μετά κατανόησα ότι ένα δίκτυο, μια διαδικτύωση θα υπάρχει για εθνικούς εισηγητές ε, από πλευράς των κρατών μελών που θα συμμετέχουν. Και η Ευρωβουλή θα έπρεπε να συμμετέχει. Είναι δυνατόν και εμείς από πλευράς μας ως εισηγητές να συμμετάσχουμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις απόψεις από πλευράς, ε, για παράδειγμα, της Σουηδικής Προεδρίας. Η κυρία Πετρίλιος αληθεύει. Πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Θα θέλετε να λάβετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν έχω να πω πολλά περισσότερα πράγματα όσον αφορά την γενικότερη προσέγγιση αυτή τη απόφαση πλαισίου. Είναι η ίδια με την προσέγγιση που έχουμε για την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Περιλαμβάνονται εδώ πέρα διατάξει για την πρόληψη, την ποινική δίωξη, διατάξει αστικού ποινικού δικαίου, αρρωγή στα θύματα και παρακολούθηση εποπτεία. Πρόκειται για μια σφαιρική προσέγγιση, πρόκειται για μια φιλόδοξη πρόταση. Ωστόσο θα ήθελα να περάσω άμεσα στα ερωτήματα που έθεσε η εισηγήτρια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς όσον αφορά την πρόληψη. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καταρχάς Στόχος μιας απόφασης πλαισίου είναι η προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Επομένω, μόνο διατάξεις οι οποίες συνδέονται στενά με το στόχο αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν και θεωρούνται ότι έχουν την κατάλληλη νομική βάση για να συμπεριληφθούν. Συντοπιώ ότι κάποιες διατάξεις για τις προλήψεις για την πρόληψη, με δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι το επίπεδο το οποίο θα θέλατε ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, αλλά νομίζω ότι η απουσία αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω άλλων δράσεων. Δεύτερον, όσον αφορά τις κυρώσεις. Θα ήθελα να πω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για το ζήτημα των κυρώσεων. Από ό,τι φαίνεται λέτε ότι το έγκλημα αυτό εφόσον διαπραχθεί εναντίον ενός παιδιού θα πρέπει να τιμωρηθεί με πάρα πολύ αυστηρή κύρωση, δηλαδή με μια ποινή που θα φτάνει τα 12 έτη. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι τα κράτη-μέλη θα είναι υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης, ενός τέτοιου υψηλού επίπεδου, μιας μέγιστης τέτοιας ποινής. Συνεπώς ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση στις επόμενες συνεδράσεις Ομάδας Εργασίας Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου. Πάντως πρέπει να σας πω ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ε, χρειαζόμαστε οι ψηλότερες, πιο αυστηρές ποινές παντού στην Ευρώπη. Το τρίτο ερώτημα είχε να κάνει με την εποπτεία, την παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής προβλέπεται μία διάταξη για την ε, δημιουργία των εθνικών εισηγητών ως σύστημα παρακολούθησης γιατί γνωρίζουμε ότι τελικά σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συλλέγονται δεδομένα προκειμένου να αξιολογούνται τα, τα πορίσματα της δράσης κατά της εμπορίας των ανθρώπων και είναι σημαντικό να υπάρχουν δεδομένα τα οποία θα είναι συγκρίσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το άτυπο τώρα δίκτυο των εθνικών εισηγητών μόλις ξεκίνησε τις δραστηριότητές του. Εξελίσσονται ακόμα συζητήσει όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων. Πάντως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όπως σας είπε η διαδικασία μόλις ξεκίνησε. Μία παρατήρηση ακόμα όσον αφορά κάποιες καινοτόμες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αρρωγή και την προστασία των θυμάτων, τη συνδρομή προς τα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει την σημαντικότητα των διατάξεων αυτών. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη, την αναγκαία υποστήριξη προς τα θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ποινικέ διαδικασίες, αλλά και στα πλαίσια της δυνατότητας απόκτησης αποζημίωσης από τα θύματα. Και γνωρίζουμε ότι ε, ο στόχος μας αυτός, το εγχείρημα μας αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά γνωρίζουμε παράλληλα ότι και τα θύματα εμπορίας είναι θύματα ενός από τα σοβαρότερα εγκλήματα που υπάρχει, που υφίστανται και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβάλλεται να προστατεύσουμε τα θύματα αυτά πάρα πολύ καλά και πολύ προσεκτικά από το πρώτο στάδιο της ποινική διαδικασίας άνευ όρων. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται και αυτό τουλάχιστον φαίνεται από την ε, ακολουθείται εθνική πρακτική ότι ε, τα θύματα θα πρέπει να προστατεύονται από την αρχή, από τα πρώτα στάδια της ποινική διαδικασίας. Εμείς αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι η αρρωγή, η συνδρομή αυτή προς τα θύματα θα δίδεται όχι μόνο στο πρώτο στάδιο, αλλά συστηματικά αυτή στιγμή αποδειχθεί ότι ένα άτομο έχει πέσει θύμα εμπορία. Και θα ήθελα εδώ πέρα να υπογραμμίσω ότι η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική διάταξη στα πλαίσια της απόφασης πλαισίου. Ευχαριστούμε πολύ εκπρόσωπο τη ε, Σουηδική προεδρία, κυρία Πετρέλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη ευρωβουλευτέ τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Υπήρχε μια ερώτηση που απευθύνθηκε προ το Συμβούλιο όσον αφορά ποινέ κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλι ε, έτυχε αναφορά. Μέσω τη ε, απόφαση ε, πλαισίου συμβαίνει το ότι οι κυρώσεις και οι ποινές έχουν διαφορετική μορφή στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Πρόκειται για ένα, όταν πρόκειται για ένα έγκλημα σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να προσαρμόζονται οι ποινές και να είναι ιδιαίτερα αυστηρές όσον αφορά ένα, μια, ένα δίκημα το οποίο έχει εγκληματική μορφή. Πρέπει να αναμείνουμε να δούμε τις διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο. Τι θα ισχύει για την ελάχιστη ποινή για ένα τέτοιο ε, έγκλημα. Όμως συμφωνούν τα κράτη-μέλη ανάμεσά τους για το ότι σοβαρά εγκλήματα, αδικήματα που έχουν ως στόχο τους παιδιά είναι τόσο σοβαρά ώστε να πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο όσον αφορά την ποινή, την κύρωση την οποία θα συνεπιφέρουν. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μεγάλη συμφωνία επ' αυτού όσον αφορά την έκθεση των παιδιών σε, τέτοια, σε τέτοιες πράξεις και πρέπει οι πράξεις να είναι αυστηρές. Παρακαλώ να είσαστε σύντομη στο χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη στο διαθέσιμο χρόνο. Η κυρία Σαρζεντίνη, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε η συγγήτρια κυρία Χέντ, Πρόκειται για καλύτερο πλαίσιο αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μα σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί ο μόνο τρόπο για να καταπολεμήσουμε την εμπορία των ανθρώπων είναι μέσω της πρόληψης και αυτό ακριβώς απουσιάζει. Επομένως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τα θύματα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λίγο πιο αυστηρό κείμενο προς αυτό και κάποιες καλύτερες πιο έξυπνες προτάσεις. Πώς μπορούμε δηλαδή να ενισχύσουμε στην πράξη τα θύματα έτσι ώστε να τους δίδεται η απαραίτητη συνδρομή όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας αλλά προκειμένου να καταφέρουν να εξασφαλίσουν και καλύτερη αποζημίωση όχι μόνο από τους υπεύθυνου του εγκλήματος, αλλά ενδεχομένως και από άλλους φορείς. Θα ήθελα ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε προ αυτό. Το σχέδιο απόφαση πλαισίου λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα τα οποία κατά την άποψή μου ποινικοποιούν το ίδιο το θύμα ακόμα περισσότερο. Λέγεται δηλαδή ότι ο πολίτης ο οποίος δέχεται υπηρεσία από άτομο που έχει πέσει θύμα εμπορίας τότε το άτομο αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί ακόμα πιο αυστηρά. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή ποινικοποιείται όμως και το ίδιο το θύμα εμπορίας και είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί στην περίπτωση αυτή ότι έχει πέσει θύμα εμπορίας. Θα μπορούσε λοιπόν το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει για ποιο λόγο βρίσκεται στην απόφαση πλαίσιο το μη δεσμευτικό αυτό άρθρο, αυτή η διάταξη και πώς μπορούν να εξασφαλίσουν στην πράξη ότι τα θύματα θα καταφέρουν να ξεφύγουν ουσιαστικά από τον κίνδυνο τη περαιτέρω ποινικοποίηση του. Εγώ νομίζω ότι η διάταξη αυτή δεν προστατεύει τα θύματα, αλλά τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα. Και όσον αφορά τα ευάλωτα και ακόμα πιο ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα. Πώς γίνεται η διάκριση αυτή. Ενδεχομένω όντω να ισχύει μια τέτοια διάκριση, αναφερθήκαμε άλλωστε σε παιδιά, αλλά θα ήθελα να πω ότι οποιοδήποτε ανθρώπινο όν το οποίο πέφτει θύμα εμπορία είναι ένα ανθρώπινο όν το οποίο είναι ευάλωτο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοια διάκριση, ιδίω όταν αυτή η διάκριση επηρεάζει την προστασία που του παρέχεται. Σα ευχαριστούμε. Μουρβάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τα τελευταία λόγια της κυρίας Αζεντίνη. Όμως θα έλεγα ότι μπορούμε με εξειδικευμένο τρόπο να έχουμε πρόληψη και υποστήριξη θυμάτων, αντίστοιχα μέτρα, αν γνωρίζουμε ποιοι είναι, ποιες είναι οι πιο συγκεκριμένα ευαίσθητες ομάδες για τις οποίες κάνουμε λόγο. Είχα ένα πρόβλημα με ένα γενικό σημείο, το σημείο 1 του 1-2 του προημείου του, της επεξήγησης, διότι κάνει λόγο για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια, τον εκπρόσωπο της εισηγήτριας, αν έγινε αυτό εσκεμένα το ότι δεν συμπεριλήφθηκε κάτι άλλο σε, αυτό το, σε αυτή τη διατύπωση. Και αυτό γιατί, διότι δεν υπάρχουν κάποια τεκμήρια για το ότι η εθνική μειονότητα θα σήμαινε ιδιαίτερα και οι γυναίκες στην περίπτωση αυτή τον Ρωμά, τον Τσιγκάνες δηλαδή. Όλοι το γνωρίζουν αυτό ότι οι Τσιγκάνες θυματοποιούνται ιδιαίτερα από τους εμπόρους, τους όσους ε, διαπράττουν το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων αν θα θέλαμε θα μπορούσαμε να είχαμε εξειδικευμένα μέτρα πρόληψης και υποστήριξης θυμάτων υπέρ αυτών των γυναικών. Εγώ όπως το βλέπω το θέμα αυτό και διαρωτώ με πάρα πολύ για τα θέματα αυτά, απασχολούμε ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα από πλευράς της ε, ε, Σουηδική Προεδρία ή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια τυφλότητα εναντί θεμάτων εθνότητα. Είναι μια, α το πούμε έτσι, ε, Υπότιτλοι ένας αποκλεισμός εθνοτικών θεμάτων. Διότι βλέπουμε τσιγκάνες γυναίκες, τσιγκάνοι εντός και εκτός της χώρας πώς αντιμετωπίζονται. Αυτό που συμβαίνει με αυτούς είναι ότι είναι θύματα μιας πολιτικής ορθότητας εντός εισαγωγικών. Γιατί, διότι εκείνοι που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα είναι και αυτοί τσιγκάνοι. Είναι οργανωμένοι εγκληματίες, μαφιόζοι, οι οποίοι κάνουν αυτό το έγκλημα, διαπράττουν αυτό το έγκλημα κατά των ε, τσιγκάνων ομοεθνών τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, θέμα εδώ που πρέπει να Θέλουμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το εθνοτικό, εθνικό στοιχείο, α το αποκαλέσω έτσι, αυτή τη εγκληματική δραστηριότητα. Μια άλλη ευάλωτη ομάδα α, είναι οι γυναίκε από τα νέα κράτη-μέλη. Γυναίκε ιδιαίτερα από τη δική μου χώρα, την Ουγγαρία. Ουγγαρέζε. δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ευαισθησία και ευάλωτου χαρακτήρα όπω οι γυναίκε από τα παλαιότερα κράτη-μέλη. Είμαστε ειλικρινεί επ' αυτού. Και για τι γυναίκε στην Ουγγαρία η κατάσταση είναι παρόμοια. Είναι παρόμοια με την κατάσταση των γυναικών από τον τρίτο κόσμο. Αν θέλουμε να κάνουμε λόγο για ένα γενικότερο πλαίσιο, να μην κάνουμε λόγο μόνο γενικά για τη φτώχεια σαν να ήταν ένα φυσικό φαινόμενο ή μια θεομηνία, αλλά να το εξειδικεύσουμε όπως και στα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες ότι σαν αποτέλεσμα διαθροτικών προσαρμογών και προγραμμάτων οικονομικής διαθροτικής προσαρμογής που μας επιβλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο οι γυναίκες καταλήγουν στη φτώχεια. Είναι λοιπόν φτωχές γυναίκες και είναι ευάλωτες και είναι, στοχοθετη... είναι ε, στοχοποιημένες θύματα αυτών των εμπόρων ε, ανθρώπων. Συγκεκριμένα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν για τις γυναίκες στα νέα ιδιαίτερα τις Ουγγαρέζες γυναίκες γυναίκες και τον εθνοτικό χαρακτήρα ιδιαίτερα των μειονοτήτων, προστατεύοντα τι τσιγκάνε γυναίκε, που είναι αντικείμενο εμπορία από του άντρε τσιγκάνου Ρωμά τη Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριο Μπουσούτιλ παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ έχω ένα ερώτημα όσον αφορά την εμπορία στα πλαίσια της παράνομης μετανάστευσης, των οδών παράνομης μετανάστευσης. Αφού του είδους η εμπορία προβλέπετε, καλύπτεται από αυτή την απόφαση πλαίσιο. Νομίζω ότι πρόκειται για τις πιο συνήθεις μορφές εμπορίας ανθρώπων που αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα στα νότια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά μιλάμε για άτομα τα οποία τα βάζουν σε μια βάρκα, του ζητάνε χίλια ευρώ ανά άτομο και τα αποστέλουν έτσι στην Ευρώπη. Αυτή η εμπορία ανθρώπων, αυτή η περίπτωση εμπορίας ανθρώπων περιλαμβάνεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής θα πρέπει να πω ότι ιδίω στα πλαίσια αυτού του είδους εμπορίες ανθρώπων έχουμε και πάρα πολλά παιδιά. Σαφώς πολλές φορές τα παιδιά αυτά συνοδεύονται από τους γονείς τους, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις ταξιδεύουν ασυνόδευτα. και καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει, ιδίω όταν μιλάμε για ευάλωτε ομάδες, που σίγουρα είναι τα παιδιά τα οποία δεν συνοδεύονται. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Χέντ, η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα μόνο. Μία απάντηση προς τα όσα είπε η κυρία Μορβάη. Εγώ ως εισηγήτρια δεν δημιούργησα αυτό το πλαίσιο απόφασης. Έτσι ούτε το συνέταξα εγώ το έχουμε μπροστά μα και το αντιμετωπίζουμε ως αντικείμενο εργασία. Όταν ιδιαίτερε εξειδικευμένε ομάδε που είναι ευάλωτε, όπω οι Τσιγκάνοι για παράδειγμα, οι Ρωμά για του οποίου έγινε λόγο από την κυρία Μορβάη, ίσω η κυρία Μορβάη μπορεί σχετικά να διατυπώσει μια τροπολογία που μπορεί να καταθέσει για να ληφθεί αυτό και να υπόψη και να καλυφθεί. Βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα τη εργασία, αντιμετωπίζοντα αυτή την απόφαση πλαίσιο. Γι' αυτό χαίρομαι και προσβλέπω στη συνεργασία και ελπίζω ότι στο τέλο θα έχουμε ένα το δυνατόν καλύτερο κείμενο. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που είσαστε και σύντομοι. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Σουηδική Προεδρία, αν επιθυμείτε να είσαστε σύντομες παρακαλώ. Ε, Θα είμαι πολύ σύντομη. Το πρώτο ερώτημα που είχε να κάνει με την ποινικοποίηση των πελατών, των χρηστών σεξουαλικών υπηρεσιών. είναι η μόνη διάταξη στην πρότασή μας που δεν είναι δεσμευτική, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε πολύ καλά το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο και γνωρίζουμε ότι σε πολλές χώρες, πολλές χώρες μάλλον κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τη διάρκεια όμως διαβούλευση που είχαμε με τα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη, είπαν με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμα να δεχθούν μια δεσμευτική διάταξη στον τομέα αυτό και γι' αυτό το λόγο ήμασταν κι εμείς πολύ προσεκτικοί γιατί θέλουμε καταρχάς να αξιολογήσουμε πρώτα την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε χώρες που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα με το ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτόν τον τομέα. Δεύτερον, ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα. Ως προς αυτό αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την διατύπωση της απόφασης πλαισίου όσον αφορά τα θύματα ποινικών διαδικασιών, όπου χρησιμοποιείται ακριβώς η φράση αυτή, ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, και για λόγους συνέπειας χρησιμοποίησαμε, επαναχρησιμοποίησαμε αυτή την ορολογία, συνειδητοποιώντας παράλληλα βέβαια ότι δημιουργείται μια σύγχυση ανάμεσα στον όρο θύματα, ευάλωτα θύματα, ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα. Και εγώ θα ήθελα να βελτιωθεί η διατύπωση αυτή στο τελικό κείμενο. Δράτω με επίσης για να σας πω ότι Εξέφρασα τι ανησυχίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προηγούμενη μου παρέμβαση, αλλά θα ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη δέχτηκαν θετικά την πρότασή μα και είχαμε μια πολύ θετική συνεργασία με τη Σουηδική Προεδρία και γενικότερα με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και πέρα από κάποια ζητήματα τα οποία θεωρούνται ακόμα αρκετά αμφιλεγόμενα, θεωρούμε ότι μια πολιτική συμφωνία θα επιτευχθεί πολύ σύντομα και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα εξωσημείωτο θετικό αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο το ευχόμαστε όλοι βέβαια, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προεδρία και κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα ζητήματα μετανάστευση, δεν καλύπτουν τα ζητήματα αυτά από την πρόταση απόφαση πλαισίου και αυτό λόγω νομική βάση. Τα ζητήματα μετανάστευση εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα, συνεπώ δεν ήταν δυνατό να συμπεριλάβουμε τα ζητήματα αυτά στην ε, τρέχουσα απόφαση πλαίσιο, η οποία είναι καθαρά κοινοτική. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με εμπορία ανθρώπων και με μετανάστευση θα αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού διαφορετικού μέσου το οποίο ενδεχομένως θα είναι μια αναθεώρηση της οδηγίας για τις άδειες διαμονής για τα θύματα εμπορίας. Αναφέρομαι στην οδηγία 81-2004. Πάντω σας επαναλαμβάνω ότι ήταν ζήτημα νομική βάση, Η Προεδρία παρακαλώ. Η ε, κυρία Πετρέλιου, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Διατυπώθηκε το ερώτημα αν αυτό το ζήτημα των ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων συζητήθηκε. Ναι, συζητήθηκε στις ε, διαβουλεύσεις, όχι μόνο για αυτό το σημείο, αλλά και σε μια διαφορετική συνάφεια. Δεν είναι κάποια, κάτι το απόλυτα καινούριο λοιπόν. Υπήρξε και μια συνεδρίαση υπό την Τσεχική Προεδρία και μια υπό την Σουηδική Προεδρία τούτο το καλοκαίρι του 2009 και αυτή η έννοια συζητήθηκε σε βάθος ευάλωτα άτομα, ευάλωτες ομάδες. Είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς ποιος και οι ποιοι είναι ιδιαίτερα, την χάνουν ιδιαίτερης ανάγκης προστασίας. Αυτό ίσως ε, μπορούσε να ε, είναι κάτι το οποίο υπενήχθηκαν και οι σημερινές διαβουλεύσεις. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Συζητήθηκε αυτό το θέμα. Και τώρα είναι θέμα της Ευρωβουλής και τώρα για τη γνωμοδότηση αυτή που έχουμε να συντάξουμε, αν υπάρχει προθυμία, αν είμαστε σε θέση να δώσουμε συνέχεια επιβάλλεται να προχωρήσουμε στο σημείο 14 τώρα, το οποίο συμπεριλαμβάνει την συνεισφορά εκπροσώπων διαφορετικών αρχών. Και έτσι σας ζητώ από πλευρά σας να είσαστε σύντομοι στη χρήση του χρόνου στις παρεμβάσεις σας. Συντομότατη, σημείο 14 λοιπόν, σύμβαση σε σχέση με την χρήση της πληροφορικής και των πληροφοριών όσον αφορά τον τελωνιακό τομέα, δηλαδή την σύμβαση CIS θα, θα γίνει παρουσίαση του εισηγητή τη Σουηδική Προεδρία, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής τη Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία των Δεδομένων, Προσωπικών Δεδομένων και τη κοινή Τελωνιακή αρχή, εποπτική Τελωνιακή αρχή. επίσης. Το, το επόμενο σημείο αφορά την αντικατάσταση της σύμβασης για την χρήση πληροφορικής για τελωνιακούς σκοπούς και πιο συγκεκριμένα θα έχουμε μια έκθεση για το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα από τον εισηγητή κύριο Αλεξάνδρ Άλβαρο πρώτα. Μετά στη συνέχεια θα γίνουν παρεμβάσεις από τη Σουηδική Προεδρία, σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της κοινή τελωνιακής αρχής εποπτικής προστασίας δεδομένων. Λοιπόν, και πάλι, σας οικετεύω, σας παρακαλώ θερμά να είσαστε συντομότατοι στις παρεμβάσεις σας. Ο κύριος Άλβαρο πρώτο, παρακαλώ. Θα σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι όσο το δυνατόν σύντομος όσο γίνεται περισσότερο. Σε αυτή τη φάση θα έλεγα ότι μπορώ να είμαι σύντομος. Πρώτα να με συγχωρήσετε για το ότι δεν ήμουν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Είχα τη χαρά να ψηφίζω στην Επιτροπή Προπολογισμών καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα σήμερα. Είμαι πισμένος τώρα ότι αγαπώ ιδιαίτερα την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο είχε ήδη παρουσιαστεί υπό την Τσεχική Προεδρία αυτό περίπου πριν από ένα εξάμεινο. Όπως προαναφέρθηκε είναι το σύστημα πληροφορικής ε, για την ενημέρωση των τελωνίων. Ο στόχος είναι αποκλειστικά να διευρυνθεί ο στόχος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα ώστε να είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την πρόληψη, την ανείχνευση και άλλα συναφή θέματα όσον αφορά ειδικά τελωνιακά θέματα και ε, ιδιομορφίες. Καταπολέμηση απατών για παράδειγμα, το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και του σεβασμού ε, των ε, διαφόρων μαρκών. Πριν από τις θερινές διακοπές σε σχέση με τα θέματα αυτά. Γνωρίζαμε ότι θα ετοίμαζε μια συνέχεια η Προεδρία. Όπως, όπως είπα δεν διέφερε και τόσο πολύ από την προηγούμενο, το προηγούμενο έγγραφο που είχε διανεμηθεί που μας δίνει μια εξοικείωση για το πώς έχουν κάποια πράγματα. Πολλά μπορούσαν, μπορεί να, μπορούν να αλλάξουν, αλλά νομίζω ότι το έγγραφο όπως έχει παρουσιαστεί είναι ένα έγγραφο επί του οποίου μπορεί να εργαστεί κανείς και να δώσει συνέχεια για το πώς έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας γνωστοποιήσω είναι ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα το σχέδιο γνωμοδότησής μας. Θα διανεμηθεί αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης στα μέλη, ώστε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης και αμέσως μετά στη συνέχεια συνέχεια άρρηκτα την επόμενη ημέρα στις 7 του μήνα Οκτωβρίου θα έχουμε συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές που είναι αρμόδιοι για τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες και ίσως όπως έχετε στο χρονδιόγραμμά σας μπορούν τροπολογίες να κατατεθούν μέχρι 12 Οκτωβρίου. Η ψήφιση ίδια θα γίνει ψηφοφορία τον Νοέμβριο. Θα έλεγα αν μπορούμε να έχουμε εντάχει διαπραγματεύσεις μετά τις συζητήσεις που ήδη είχαμε με τη Σουηδική Προεδρία σε άτυπο επίπεδο μπορούμε έτσι να ολοκληρώσουμε εισαγωγικών να το πω έτσι το χαρτοφυλάκιο φύση όλων και έγκαιρα ιδιαίτερα παραμένοντας μέσα στο πλαίσιο της Σουηδικής Προεδρίας, διότι γνωρίζω ότι θέλουν να ολοκληρώσουν αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτή την πτυχή. Ουσιαστικά θα έχουμε συζητήσεις και προσκαλώ τους ισχυώδεις εισηγητές να το κάνουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα που πρέπει να δούμε είναι πώς κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Θα με ενδιαφέρει βέβαια να ακούσω την άποψη της ε, Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για την διατύπωση που διανεμήθηκε και είναι επίσημο κείμενο ή διανεμήθηκε υστερότερα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά το εύρος της οδηγίας, θέματα πρόσβασης, ε, προσπελασιμότητας. Παρότι αναφέρονται κάποια πράγματα στο έγγραφο που έχουμε στα χαρτιά μας, κάποιες εξειδικεύσεις και διευκρινήσεις, αποσαφηνήσεις μπορούν να δοθούν. Με μια πρώτη ματιά υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις μεταξύ διαφορετικών άρθρων που θα προσπαθούσαμε να περιορίσουμε αν είναι δυνατόν και να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και κανόνες. Τεχνικά, από τεχνική πλευρά είναι κάτι που θα θέλαμε να μπορέσουμε να πετύχουμε μέσα στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχουν ίσως κάποια θέματα που αφορούν τη διαφάνεια. Ήδη έχουμε δει κάποια θέματα και με που θα μπορούσαν να καλύψουν τέτοιες περιπτώσεις. Όμως ουσιαστικά θα έπρεπε κανείς να δώσει να αξιολογήσει θετικά τις επιδόσεις της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Βελτίωσαν το έγγραφο σε σχέση με τη διατύπωση των Γάλλων της Γαλλικής Προεδρίας και μετά των Τσέχων. Αυτό που βλέπουμε τώρα δείχνει ότι υπήρξαν εξελίξεις στο Συμβούλιο, έλαβαν υπόψη σε κάποιες περιπτώσεις κάποια πράγματα, υπήρξαν βελτιώσεις, ελήφθησαν υπόψη οι απόψει του Κοινοβουλίου πριν από τις θερινές διακοπές Σημειώνεται θετική πρόοδος λοιπόν και νομίζω έγκαιρα θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σεβόμενοι τις προδιαγραφές, τις προθεσμίες μέσα στο χρονοδιάγραμμα και να ψηφίσουμε κατά τα τέλη Νοεμβρίου στην Ολομέλεια και μέχρι τότε όπως είπα θα κληθούν οι σκιώδεις εισηγητές να γνωμοδοτήσουν όταν θα έχει οριμάσει, θα είναι έτοιμη ε, η γνωμοδότηση, ο σχέδιο γνωμοδότησης και μέσα στις προθεσμίες θα καταφέρουμε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια να ολοκληρώσουμε στην πρώτη ανάγνωση αν γίνεται. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και τη υπηρεσία Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ποιες είναι οι συστάσεις τους σε σχέση με το έχουν διαμορφωθεί τώρα τα πράγματα. Και πάλι πρέπει να συγχαρώ τη Σουηδική Προεδρία για άλλη μια φορά, διότι βελτίωσε αυτό το έγγραφο σε σχέση με αυτά που είχαμε ω αρχικό έγγραφο στα χέρια μα στο παρελθόν. Νομίζω υπαρκούν αυτά για τώρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Άλβαρο. Εξ ονόματο Προεδρία, η κυρία Κάλμ, για ένα δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσαμε και πριν από λίγο, οι συζητήσεις ξεκίνησαν στην αρμόδια ομάδα εργασίας Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2008 μετά από πρόταση της Γαλλίας. Όπως επίσης ακούσαμε, ήδη υπάρχει μία σύμβαση που καλύπτει τα συστήματα πληροφορικής των τελωνίων, η οποία υπάρχει από το 1995. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να αναθεωρήσουμε τη νομική βάση για το σύστημα αυτό. Η βασική ιδέα της αναθεώρησης ήταν να ασχοληθούμε με τον κανονισμό 415 του 1997 που είναι ο κανονισμός που εμπίπτει στον πρώτο πυλώνα και να κάνουμε τι απαραίτητε εκεί τροποποιήσει. Καθώ επίση και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι διάφορε υπηρεσίε εφαρμογή του κανονισμού αυτού στα κράτη-μέλη. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κανονισμό αυτό προκειμένου να συνάδει πλέον με όλες τις διατάξεις που βρίσκονται στον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και πιστεύουμε τόσο το Συμβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ σημαντικό να προβλέπεται μια πλήρη προστασία της ακαιρεότητας των ανθρώπων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με την επικαιροποίηση αυτή των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων έχουμε πετύχει το στόχο αυτό. Επίσης, δίνουμε πλέον την ε, δυνατότητα σε εθνικές αρχές να καταχωρούν πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για στρατηγική ανάλυση και όχι μόνο για απλούς ελέγχους και επιτήρηση όπως γινόταν στο παρελθόν. Επίσης, δημιουργούμε τη δυνατότητα για την Ευρωπόλ και τη Eurojust να έχουν πρόσβαση στο σύστημα αυτό σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη δική τους εντολή βέβαια. Έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν πληροφορίες στο σύστημα κάτι που στο παρελθόν ίσχυε μόνο για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να συνοψίσω και για να μην μακρηγορήσω και πολύ, θα ήθελα να σας παρουσιάσω πολύ γρήγορα πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Ολοκληρώσαμε την τεχνική ενάγνωση του κειμένου στην αρμόδια ομάδα εργασία του Συμβουλίου και κρεμούν δύο ζητήματα αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να επιλύσουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την πρόσβαση στο σύστημα από τη Eurojust. Το αν δηλαδή η Eurojust θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο σύνολο του συστήματος, σε όλο δηλαδή το σύστημα, δηλαδή και στις δύο βάσεις δεδομένων, η μία έχει να κάνει με την εποπτεία και η άλλη έχει να κάνει με την καταχώρηση πληροφοριών, όσον αφορά τις τρέχουσες και ολοκληρωμένε έρευνες. Και το δεύτερο ζήτημα το οποίο εκκρεμεί είναι ποιος θα πρέπει να είναι ο αρμόδιος για την εποπτεία του συστήματος. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα δούμε και ποιο ενδιαφέρεται για τη θέση αυτή. Ελπίζουμε ότι τα δύο αυτά κρεμή ζητήματα θα επιληθούν και ότι θα καταφέρουμε έτσι να υιοθετήσουμε το σχέδιο κειμένου και να καταλήξουμε έτσι σε μια νέα απόφαση του Συμβουλίου, αναθεωρημένη πλέον. Ολοκληρώνοντα, να σα πω ότι είμαι στη διάθεσή σα για ενδεχόμενε ερωτήσει, παρατηρήσει σα. Έχουμε ήδη λάβει κάποιε παρατηρήσει από εσά και θα προσπαθήσουμε να τι λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, διορθώνει ο πρόεδρο, τον κύριο Τιερή, ένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την υποστήριξη της Κομισιόν στο κείμενο του Συμβουλίου διότι είναι απαραίτητο να εξεταστούν παράλληλα οι διατάξεις αμοιβαία συνεργασίας του πρώτου πυλώνα με εκείνες της διοικητικής συνεργασίας του τρίτου. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα στη συνεργασία μεταξύ Europol και Eurojust και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα του προϋπολογισμού. Η Κομισιόν αντιμετωπίζει δύο-τρεις ε, μίζωνες ε, δυσκολίες όπου η Κομισιόν θα ήθελε το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στις τράπεζες δεδομένων ε, της Eurojust και της Europol. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι για την προστασία των δεδομένων ε, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της EPS και των Εθνικών Υπηρεσιών Προστασίας Δεδομένων. Αν σε αυτό το πλέγμα περιφρούρησης προσθέσουμε και την GCE ε, τότε επιβαρύνεται ιδιαίτερα το σύστημα και δυσλειτουργεί. και ξεφεύγουμε από το ευρωπαϊκό μοντέλο προστασίας των δεδομένων έτσι όπως προβλέπεται στον τρίτο πυλώνα. Την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε ότι ο προϋπολογισμός μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή 20% μείωση, οπότε δύσκολα μπορούμε να εφαρμόσουμε το νέο σύστημα. Πόσο μάλλον που έχουμε και σημαντικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να αναλυφθούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλω να επιστήσω επίσης την προσοχή του σώματος στο ότι περνάει από ό,τι φαίνεται η μείωση αυτή του ενός εκατομμυρίου από το Συμβούλιο και αυτό μας δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και θέλουμε να το έχετε υπόψη σας. Ο κύριος Ζωβάνι Μπουταρέλη από την Επιτροπή Προστασία, από τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Είχα έρθει και στα τέλη Μαρτίου, θυμάστε, σε μια ακρόαση. Μετά την ακρόαση αυτή, η EDPS ενέκρινε τον ε, Απρίλιο μία λεπτομερή γνωμοδότηση σε σχέση με την πρόταση αυτή την οποία συζητάμε. Δεν θα ήθελα να εκθέσω τώρα όλα τα επιχειρήματα τη γνωμοδότηση αυτή από την Ευρωπαίου Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ε, εργασία που έχει κάνει τόσο ο συγητή Αλβάρο όσο και η Σουδική Προεδρία. Θα ήθελα να τονίσω ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την εποπτεία. Η EDPS είναι υπέρ της ε, έγκρισης του ίδιου μοντέλου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υποστηρίξει για το σύστημα SIS, Schengen Information System 2, και για το σύστημα το οποίο ακολουθείται για τις ευρωπαϊκές αγορές και για τη Eurodac. Το μοντέλο αυτό συνάδει με τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της ε, Επιτροπής προστασίας δεδομένων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο μοντέλο. Στόχος της γαλλικής πρωτοβουλίας είναι να ευθυγραμμιστεί το τμήμα του, το, του τρίτου πυλώνα με το τμήμα εκείνο του πρώτου πυλώνα και να δημιουργηθεί ένα πιο ενιαίο σύστημα. Κατά την άποψή μας η ευθυγράμμιση αυτή θα πρέπει να γίνει και στην εποπτεία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι θα υπάρχει μία εξωτερική συνέπεια του συστήματος αυτού με άλλα ανάλογα σύστημα όπου υπάρχει ένα συντονισμένο σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας τόσο για τα τμήματα του πρώτου και για τα τμήματα του τρίτου πυλώνα. Και αυτό ήδη ισχύει εδώ και κάποια χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα σε άλλα συστήματα. Τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα, παρόμοιες προκλήσεις όσον αφορά την εποπτεία. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια εσωτερική συνέπεια ανάμεσα στο πρώτο και το τρίτο πυλώνα για τα ζητήματα που άπτονται των ε, τελωνίων. Ξέρετε ότι ο EDPS είναι ουσιαστικά Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων για το τμήμα του πρώτου πυλώνα του συστήματος και μετά την δεύτερη γνωμοδότηση την, ε, της Ομάδας Εργασίας για τη Τελωνία του Ιουλίου εξακολουθούμε να πιστεύουμε Μετά τη γνωμοδότηση με συγχωρείτε των Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό και μία ευθυγραμμισμένη εποπτεία. Το ευθυγραμμισμένο αυτό μοντέλο δεν θα αποδυναμώσει καθόλου τις εθνικές αρχές. Θα συνεχίσουν οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο που διαδραματίζουν μέχρι τώρα. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αυτές αρχές θα συντονιστούν ε, στις Βρυξέλλες. Θα καταφέρουν δηλαδή να έχουν ένα μια συντονισμένη προσέγγιση ή να ευθυγραμμιστούν και να συντονιστούν στα πλαίσια ενός ενιαίου οργάνου όπως το CJSA. Πέρα από τα ζητήματα αυτά της νομικής συνοχής και διαφάνειας, πιστεύουμε ότι το μοντέλο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί και για πρακτικούς λόγους και για λόγους εξοικονόμησης. Σκεφτείτε απλώς τις, το, πόσες συνεδριάσεις χρειάστηκε να κάνουμε προκειμένου να διοργανώσουμε τις συνεδριάσεις αυτές που γίνονται δύο φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες. Όλο αυτό το σύστημα συνεδριάσεων θα εξορθολογηθεί. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα καλύτερο επίπεδο διαφάνειας θα καταφέρουμε να αποφύγουμε το να έχουμε δύο συστήματα εποπτεία στα πλαίσια ενό κοινού συστήματο, πράγμα το οποίο είναι δικαιολόγητο. Με την GSA, την Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή επαφή, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Δεν υπάρχει απόκληση όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν απλώς κάποιες αποκλήσεις όσον αφορά τις μελλοντικέ προοπτικές. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες και σας ζητούμε να ακολουθηθεί ένα παρόμοιο μοντέλο εποπτείας στο ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε για την Τελωνία με αυτό το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ήδη στη Eurodac και με αυτό το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για τον πρώτο πυλώνα του ΣΥΣ. Επίσης το επιχείρημα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε εντελώ διαφορετικές βάσεις δεδομένων στους δύο πυλώνες που εξυπηρετούν εντελώ διαφορετικού σκοπού και δεν συνδέονται μεταξύ του, δεν είναι πιστικό το επιχείρημα αυτό. Εμεί θεωρούμε ότι στην πράξη έχουμε δημιουργήσει μία τεχνική διάκριση ανάμεσα στους δύο αυτούς πυλώνες και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και λίγο το μέλλον, δηλαδή την θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τα δύο αυτά παράλληλα μοντέλα εποπτείας σε ένα νέο καθεστώς το οποίο δεν θα εφίστανται πλέον πυλώνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαστε στη θέση σας για περισσότερες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα εξ ονόματος της κοινή εποπτικής αρχής των τελωνίων θα λάβει τον λόγο ο κύριος Πίτερ Μάικρο. Τρία λεπτά κατά το μέγιστο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε τρία λεπτά να ολοκληρώσω. Εκπροσωπώ την κοινή τελωνιακή αρχή εποπτείας, όπου όλες οι ανεξάρτητες αρχές των 27 κρατών μελών συνεργάζονται σε αυτήν. Δεν μπορώ να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες απαντώντας σε θέματα που προαναφέρθηκαν. Όμως το ζήτημα, το κύριο ζήτημα είναι ότι η δουλειά από πλευράς των οργανισμών τελωνίων βασίζεται σε μια απόφαση πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην επιβολή του δικαίου. Τονίζει ιδιαίτερα την εθνική εποπτεία αυτή η απόφαση. Αν αξιολογήσει κανείς αν το σύστημα πληροφοριών για τα τελωνία στην επιβολή του νόμου και τα αξιολογήσει κανείς, θα δει κανείς ότι είναι με συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, με τεχνικές δυνατότητες και ε, δυνατότητες διευκόλυνσης που παρέχονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό ήταν ο λόγος γιατί όλες οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτού του είδους η εργασία, αυτό το έργο σε σχέση με το Schengen Information System και το Visa Information System θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για την θεσμοποιημένη αυτή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, διότι είναι αυτή η δουλειά τους. Και μια και πρέπει να υποπτεύουν τη συμμόρφωση με την απόφαση πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η περισσότερη δουλειά συσχετίζεται άμεσα με το τι γίνεται στα ίδια τα κράτη-μέλη και όχι με το τι τεκταίνεται εδώ στις Βρυξέλλες από πλευρά συστηματι... προσέγγισης όσον αφορά το σύστημα. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο οι εθνικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα να διατηρηθεί αυτή η κοινή εποπτική αρχή. Πράγμα το οποίο δεν εκπλήσει, διότι και η Eurojust έχει μια αντίστοιχη διάρθρωση, μια αντίστοιχη δομή και η Euro το ίδιο και έτσι είναι η καλύτερη οδός να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται η εποπτεία θα έχει επίπτωση και στο εθνικό επίπεδο. Είναι οι εθνικές αρχές εποπτείας που μπορούν να, αποκοινούν να καταλήξουν στο επίπεδο ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό διασφαλίζει και δημιουργεί δυνατότητα καλύτερη συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. Λογικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ του EDPS και με το EDPS να υπάρχει συνεργασία σε σχέση όσον αφορά τις εποπτικές αρχές. Αυτή η λογική προσέγγιση είναι μέρος της συνολικής προσέγγισης, ότι το τμήμα ασφάλειας που αφορά την ασφάλεια αυτού του συστήματος που αποτελεί τμήμα των εργασιών πρέπει να γίνεται μέσα στο πλαίσιο της EDPS. Λοιπόν, συνεργασία και πάλι συνεργασία από την άλλη πλευρά με την κοινή εποπτική αρχή όπου συνεργάζονται οι εθνικές αρχές εποπτείας προς την ευόδοση του στόχου. Άκουσα τον λόγο Ευρωπαϊκή Προστασία προσωπικών δεδομένων. Αλλά δεν ε, γνωρίζω καμιά συζήτηση είτε στην Ευρωβουλή είτε στο δικό μας πλαίσιο είτε μεταξύ των εθνικών εκπροσώπων εποπτείας για κάτι τέτοιο. Μια όμως και γίνεται χρήση αυτού του όρου γίνεται χρήση για κάτι το οποίο δεν υφίσταται, για κάτι το ανύπαρκτο. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο οι εθνικέ αρχέ διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων στρεφόμενε προ το μέλλον για να δουν το τι θα γίνει μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα ήδη συμμετέχουν σε διάφορα φόρα για να συζητήσουν πώ θα διασφαλιστεί η προστασία προσωπικών δεδομένων μετά την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα και την αλλαγή των νομικών διαρθρώσεων ώστε να προστατεύονται με τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά τον λόγο κανένα άλλο. Ίσως είναι ο χρόνος να αντιδράσει τώρα και να τοποθετηθεί ο κύριος Άλβαρος, εισηγητής. Α, ένα, δευτερο, ένα λεπτό. Φαίνεται ότι κάποια ερώτηση υπάρχει. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ παίρνω το λόγο ως και όδηση εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω τον πρόσωπο της Σουηδικής Προεδρίας όπως και τον εισηγητή για την εργασία τους. Και θα ήθελα να πω ότι το πρώτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η προστασία των δεδομένων. Είναι σημαντικότατο να παραμείνουν μυστικά αυτά τα στοιχεία υπό την κυδαιμονία των αρμοδίων αρχών. Θα πρέπει να δούμε επίσης ποια θα είναι η εποπτική αρχή. Σίγουρα θα έχουμε μία καρποφόρα συνεργασία με τον εισηγητή. Θα πρέπει να σκεφτούμε ακόμη περισσότερο τα κείμενα για τον τρόπο προστασίας των δεδομένων και θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τη συζήτηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να αποφασιστούν. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιώτοβα. Τώρα θα λάβει τον λόγο και πάλι ο κύριος Άλβαρο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης και την κυρία Γιώτοβα. Ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά της. Την ευχαριστώ για την υποστήριξη, την υποστήριξη της ομάδας S&D. S&D. Είμαστε πάντα ιδιαίτερα ευτυχείς όταν υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Τώρα, ενδιαφέρον θα είναι πώς το Συμβούλιο θα επιλύσει το πρόβλημα σε σχέση με το, αυτά που έγιναν από τη Eurojust. Προσωπικά, σκεπτόμενοι γι' αυτό, η πρώτη πρόθεση ήταν, η αρχική πρόθεση, και γι' αυτό με ενδιαφέρει να δω την τελική λύση από το Συμβούλιο. Ουσιαστικά θα έχουμε δύο διαφορετικά καθεστώτα, μια και η Europol και η Eurojust έχουν διαφορετικά καθήκοντα και μεταξύ τους και οι δύο έχουν διαφορετικά καθεστώτα. Λοιπόν, θα είχε νόημα να το δούμε αυτό, όμως προσβλέπω να δω τι θα γίνει σε σχέση με την τελική ρύθμιση. Όταν έχουμε την εποπτεία του συστήματος, συμφωνώ με τον επόπτη των προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια και έχουμε μια πρακτική, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν, να αλλάξουν αυτά τα πράγματα με το ε, σύστημα ε, πληροφορικής για τα τελωνία. Ουσιαστικά λειτουργεί καλά και καθότι βλέπω η δομή για την εναλλακτική δυνατότητα 1, δηλαδή να υπάρξει μία αρχή με δύο εκπροσώπους από κάθε κράτος μέλος, δηλαδή θα καταλήγαμε σε κάτι σαν την γερουσία στη ΣΥΠΑ και θα ήταν αρμόδια αυτή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 54 μέλη, 2 επί 27 ίσον 54. Δύο εκπρόσωποι από κάθε κράτος μέλος δηλαδή. Και αν λάβουμε υπόψη και άλλα θεσμικά όργανα που θα ήθελαν να εμπλακούν και να συμμετάσχουν, δεν ξέρω 100% πως όλα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά. Υπάρχει λοιπόν, ας το πω, πώς να το πω, σε σχέση με ένα δεδομένο πρότυπο μια και δεν είναι δεδομένο κάτι τέτοιο έχουμε το 2058 ε, την, τις οδηγίες ε, υπάρχει ας το πω έτσι μέσω πρακτικής εφαρμογής και εκπείρας ένα πρότυπο για το τι κάνουμε με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με συνέπεια εργάστηκε η Ευρωβουλή για να δει αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα με τελικό το πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων απόφαση πλαίσιο του 2008. Θεωρούσαμε πάντα ως Ευρωβουλή ότι ο επόπτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο για αυτά τα θέματα συμπληρωματικά σε σχέση με το άρθρο 29 και την ομάδα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 που καλύπτει τα περισσότερα από τα συναφή αυτά θέματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ ίσως θα υπήρχε κάποια προτίμηση αλλά τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να αναφερθώ για το ποιο πρότυπο θα ε, επιλέγαμε. Όμως ακούσαμε επίσης και τις ανησυχίες για τον περιορισμό κατά ένα εκατομμύριο ή σε ένα εκατομμύριο. Δεν είναι αυτό ουσιαστικά το θέμα που εξετάζουμε. Είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών που επιφορτίζεται με τέτοια θέματα. Και μια και ανήκω και στις δύο, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, δηλαδή, να δούμε επίσης για να καθησυχάσω τις ανησυχίες κάποιων, οι πληρωμές είναι οι ίδιες. 4,5 εκατομμύρια πληρωμές. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό το οποίο μειώθηκε, μειώθηκε και ήταν το 1 εκατομμύριο που αναφέρθηκε, ήταν οι υποχρεώσεις από 6,5 ε, εκατομμύρια είχαμε 5,5 εκατομμύρια στις υποχρεώσεις. Όμως οι πληρωμές δεν αλλάζουν, αυτές παραμένουν σε 4,5 εκατομμύρια και αυτό πρέπει να δούμε υπό τους όρους χρηματοδότησης. Όμως τούτων λεχθέντων παρόλα αυτά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι άκουσα ότι και το EDPS και τα θεσμικά όργανα είναι πρόθυμα να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα υπάρξει αναφορά. Όπως είπα, την επόμενη εβδομάδα μετά την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης θα συναντηθούμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Θα υπάρχει περίοδος πέντε ημερών για τη διατύπωση τροπολογιών. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ε, συμφωνήσουν μαζί μου σε αυτή τη διαδικασία, να είναι ταχεία η διαδικασία και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και όταν θα γίνει αυτό υπάρχει αρκετό πλαίσιο, αρκετό περιθώριο να συζητήσουμε με τις αρχές και τα θεσμικά όργανα που θα εμπλέκονται, να βρούμε μια ταχεία και ορθή λύση ποιε δυνατότητες θα δοθούν από πλευράς ρυθμίσεων. Τώρα, σε σχέση με τη δική μας Επιτροπή δεν νομίζω ότι σε σχέση με εμάς αυτό είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο δημιουργεί τριβές ή πιέσεις. Ευχαριστώ έχουν αναφερθεί τα θέματα αυτά και ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης διαδικαστικά και μπορούμε να συνεχίσουμε δίνοντας, ε, να συνεχίσουμε στο μέλλον σχετικά. Περνάμε στην ευθεία γραμμή, τελική ευθεία της σημερινής μας συνεδρίασης ε, απόψε. Τελικό σημείο, τελευταίο σημείο είναι το 15 για απόψε. Διαπίστευση των ε, δραστηριοτήτων εγκληματολογικών εργαστηρίων, ιατροδικαστικών εργαστηρίων. Ο εισηγητής συντάκτης αυτού, αυτής της έκθεσης είναι ο κ. Τίμωθη Κέκοπ. Είναι όμως φοβούμε δεν απουσιάζει αυτή τη στιγμή, δεν παρίσταται και όλοι γνωρίζουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και που αφορά προσωπικά στοιχεία της προσωπικής ζωής, ζωής όπως το προφίλ DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα τέτοια προσωπικά στοιχεία και η διαπίστευση των εγκληματολογικών εργαστηρίων και διεργασιών είναι σημαντικό βήμα προς την ανταλλαγή αυτών των επιστημονικών στοιχείων σε ένα ασφαλέστερο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καλύτερος τρόπος να, ακούς, να προχωρήσουμε είναι να μας μιλήσει πρώτα η Σουηδική Προεδρία, μετά ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα έχουμε και χρόνο για τη συζήτηση. Σουηδική Προεδρία λοιπόν πρώτα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να σας παρουσιάσω μία σουηδική και ισπανική πρόταση για μία απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την διαπίστευση για τις διαδικασίες των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Παρουσιάσαμε την πρόταση αυτή τον Ιούνιο του 2009 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει μέχρι, μέχρι την 26 Νοεμβρίου. Στόχος της πρότασης αυτής είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των δεδομένων εκείνων που διακινούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη καταρχάς των πολιτών μας, ότι μπορούν δηλαδή να βασίζονται στην ποιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τις διοκτικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη είναι της ίδιας ποιότητας με τα δεδομένα που έχουν οι αρχές αυτές και χρησιμοποιούν σε εθνικό επίπεδο. Η ανάγκη λοιπόν αυτή για κοινά ποιοτικά πρότυπα αναγνωρίστηκε και σε προηγούμενα κείμενα του Συμβουλίου και θα ήθελα να σπαραπέψω στο πρόγραμμα της Χάγης καθώς επίσης και στην απόφαση του Συμβουλίου για την εφαρμογή του ΠΡΟΥΝ. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αγνοούμε το ότι ε, πολλές φορές δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα σε διάφορα εργαστήρια, σε διάφορα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζετε, το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι σε πολύ μεγα... μάλλον ανταλλάσσονται ήδη σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο όμως για τον τελικό χρήστη να αξιολογήσει την ποιότητα των δεδομένων αυτών. Ακόμα και αν ένα κράτος μέλος ισχυριστεί ότι έχει στα χέρια του δεδομένα πολύ ψηλής ποιότητος, αυτό δεν σημαίνει σπουδαία πράγματα για έναν εμπειρογνώμονα από ένα άλλο κράτο μέλο. Γιατί ενδεχομένω πάντα να υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν θα έχουν διευκρινιστεί, αν η αποθήκευση των δεδομένων έχει γίνει σωστά, αν η καταχώρηση των δεδομένων έχει γίνει σωστά, από τη στιγμή που φτάνει στο εργαστήριο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Προκειμένου λοιπόν να αξιολογηθεί η ποιότητα ενό εργαστηρίου, θέλουμε να γνωρίζουμε αν τα εργαστήρια σε τακτική βάση αξιολογούν τις ικανότητες των εργαζομένων τους και είναι πολύ σημαντικό επίσης και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της ανάλυσης από τα εργαστήρια αυτά να είναι επίκαιρος, να είναι σύγχρονος, να τυχαίνει της κατάλληλης συντήρησης. Χωρίς λοιπόν την πιστοποίηση πάντα θα υπάρχουν τα ερωτήματα αυτά και δεν θα γνωρίζουμε τελικά ποια, ποιο δρόμο έχει ακολουθήσει το δεδομένο από τη στιγμή που έφτασε σε ένα εργαστήριο και από τη στιγμή που α, ανταλλάσσεται με ένα άλλο κράτος μέλος ή που ερμηνεύεται με τον αβ τρόπο στα πλαίσια μιας μελέτης. Έτσι λοιπόν, τα απορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων θα πρέπει να είναι αξιόπιστα ανεξάρτητα από το που βρίσκεται το εγκληματολογικό αυτοεργαστήριο οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξασφαλίζοντα λοιπόν ότι όλα τα εργαστήρια θα είναι διαπιστευμένα χρησιμοποιώντας τα ίδια διεθνή κριτήρια ISO 7825, ISO 7825, θα καταφέρουμε δηλαδή να διευκολύνουμε τους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα είναι σε θέση να εξελογούν καλύτερα την ποιότητα των πορισμάτων που χρησιμοποιούν. Των πορισμάτων δηλαδή που απορρέουν από κλιματολογικά εργαστήρια. Θα πιστοποιείτε δηλαδή ότι όντω είναι εγκληματολογικό εργαστήριο πλήρη διεθνή πρότυπα ποιότητο. Το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση αυτή περιορίζεται καταρχά στα δακτυλικά αποτυπώματα και στο DNA. Θα γνωρίζετε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA είναι πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για τις διοκτικές αρχές. Είναι πολύ αποτελεσματικά γιατί βοηθούν τις τοπικές αρχές να ταυτοποιήσουν ύποπτους και χρησιμοποιούνται επίσης και για την απελευθέρωση αθώων κρατούμενων. Το πεδίο φορμαγής επίσης έχει περιοριστεί στις δραστηριότητες των εργαστηρίων. Δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση αυτή καθόλου ο χώρος, ο τόπος του εγκλήματος. Όσον αφορά τώρα το πρότυπο αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το Διεθνές Αυτοπρότυπο 1725 για τις ε, εγκληματολογικές ε, ε, συγγνώμη, για διαδικασίες των εγκληματολογικών εργαστηρίων περιλαμβάνει δύο βασικές απαιτήσεις. Πρώτον, management requirements, απαιτήσει που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, το management ενός εργαστηρίου και δεύτερον, εν, κάποια τεχνικά κριτήρια, τεχνικές απαιτήσει όσον αφορά την επάρκεια των εργαζομένων, καθώς επίσης και την επάρκεια του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε όντως την συνολική επάρκεια ενός εργαστηρίου. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι με την πρόταση αυτή δεν πρόκειται να ευθυγραμμίσουμε τους, τις μεθόδους που ακολουθούνται. Το πρότυπο αυτό δεν υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Το μόνο το οποίο λέει το πρότυπο αυτό είναι ότι οποιαδήποτε μέθος χρησιμοποιεί ένα κλιματολογικό εργαστήριο θα πρέπει η μέθοδος αυτή να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια. Καταλήγουμε έτσι στην, σε εγκληματολογικά εργαστήρια τα οποία θα είναι επιστοποιημένα, τα οποία θα χρησιμοποιούν μεθόδους και μέσα τα οποία θα είναι αναγνωρισμένα. Και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι τα πορίσματα και η ανάλυση των εργαστηρίων αυτών είναι ποιοτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες. Αυτά όσον αφορά μια σύντομη παρουσίαση της πρότασης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα θέλαμε να γνωρίσουμε και ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ρενέ Βαντέκ, παρακαλώ. Σε τρία λεπτά παρακαλώ, κατά πολύ. Αυτό θα βοηθούσε όλους μας να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Θα είμαι το δυνατόν σύντομος. Χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρωτοβουλία για την διαπίστευση εγκληματολογικών τέτοιων δεδομένων και δραστηριοτήτων όταν ε, υπάρχει διαπίστευση σε αυτά τα εργαστήρια και προσαρμοζόμαστε στις διεθνείς προδιαγραφές, ε, εγγυόμαστε την ποιότητα του έργου αυτών των πειραματικών ε, εργαστηρίων στα κράτη-μέλη. Και αυτό δημιουργεί αμοιβή εμπιστοσύνη για τα αποτελέσματά τους όταν τα αποτελέσματα όσον αφορά το DNA για παράδειγμα είναι διαπιστευμένα θα είναι εξίσου αξιόπιστα όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Οι πιθανότητε σφαλμάτων όσον αφορά τι διεργασίε στα πειραματικά εργαστήρια μπορούν να μειωθούν και σαν αποτέλεσμα οι ευκαιρίε να εμπλακούν κάποιοι άδικα ε, στην δίωξη μειώνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θετικό αποτέλεσμα. Θα παρακολουθήσει τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεισφέρει όπου είναι δυνατόν θετικά και ελπίζω ότι ήμουν αρκετά σύντομος, Πρόεδρε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τον λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που συνεργαστήκατε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Φαντεν Κάπ έχει τον λόγο τώρα. Όχι. Τζάκι Φώστερ. Τζάκι Φώστερ. Εξ ονόματος. Ναι, παρακαλώ. Εσείς έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Και να ζητήσω συγγνώμη για τον κύριο Κέρκοπ που είναι ο εισηγητής που δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και απουσιάζει. Φυσικά είδαμε το έγγραφο του Συμβουλίου και φυσικά και άλλα έγγραφα. Και έτσι θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα που ίσως δεν θα είναι δυνατόν να απαντηθούν απόψε αλλά νομίζω ότι θα ήταν επικοδομητικές ερωτήσεις για την, τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής και πρέπει να απαντηθούν. Ως θέμα αρχής θα υποστηρίζαμε μέτρα να υπάρξει καταστολή εγκληματικών δραστηριοτήτων και αυτό ισχύει ε, σε πλήρες μέτρο για όλα τα θέματα. Τώρα για το DNA και άλλα συναφή. Νομίζω πιθανώς θα γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα όταν βλέπουμε συλλογή δεδομένων DNA ανά κράτος μέλος, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που ισχύουν από κράτος σε κράτος και σε εθνικό επίπεδο αυτό για την συλλογή και αποθήκευση του DNA. Είναι λοιπόν κάτι που πρέπει πάντα να θυμόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι απλό το πράγμα. Γιατί κάνουμε λόγο εδώ για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για άλλα συναφή. Μην πιστεύει κανείς ότι είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Αυτό όσο αφορά την, την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων επίσης και πάλι. Για τα έγγραφα τα οποία έχετε ε, ετοιμάσει θα ήθελα να ερωτήσω τα εξής Θεωρούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη, θεωρείται ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη οδηγία. Ερώτηση, μπορείτε να μας δώσετε κάποια άποψη. Πόσα κράτη-μέλη ήδη συμμορφώνονται με αυτές τις προδιαγραφές. Σε ένα αρχικό έγγραφο Είπατε ότι είχε αποσταλεί ένα ερωτηματολόγιο για το πώς έχουν τα πράγματα από κράτος σε κράτος. Αυτές οι πληροφορίες αυτών των ερωτηματολογίων θα ήταν πολύ χρήσιμες για τα μέλη της Επιτροπής μας, διότι δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου σας. Επιπρόσθετα είπατε ότι θα γινόταν σεμινάριο στη Στοχόλμη 2 και 3 Ιουνίου. Ερώτηση, προχώρησε η διεξαγωγή αυτού του σεμιναρίου και ποια ήταν η έκβασή του και το αποτέλεσμα αυτού. Στη συνέχεια, είχατε πει επίσης ότι είχατε μια ομάδα εργασία, λέει, που θα συνερχόταν υπό τη Σουηδική Προεδρία. Θα θέλαμε να μάθουμε, συνήλθε αυτή η ομάδα εργασία. Και σε σχέση και με το σεμινάριο, κάτι φαίνεται ότι ε, ίσω υπήρχε στο έγγραφό σα. Επίση, ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει λύσει ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την συγχρηματοδότηση αυτών των μέτρων. Τι ακριβώ σημαίνει αυτό το θέμα συγχρηματοδότηση και τι σημαίνει και το θέμα τη επαναχρηματοδότηση, που αυτό το θέμα θα τεθεί σίγουρα και πρέπει να απαντηθεί. Θέλατε στενότερη συνεργασία με το δίκτυο των εγκληματολογικών ε, ιδρυμάτων. Συνεργασία και για την διαπίστευση. Πώς βλέπετε ότι μπορεί να σφυριλατηθεί και να διατηρηθεί αυτή η συνεργασία, να προαχθεί και να ευδοκιμήσει. Τελική παρατήρηση. Ποιος ακριβώς θα αποφασίσει για τα θέματα και μεθόδους διαπίστευσης. Υπάρχουν λοιπόν σίγουρα ερωτήσεις εδώ που εσείς τονίσατε στις πτυχές του εγγράφου σας, αλλά δεν είχαμε τη χαρά ακόμα να δοθούν απαντήσεις επ' αυτών τελεσίδικε. Και επίση θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω κανεί να είναι εναντίον τη αμοιβαία αναγνώριση και διαπίστευση. Είναι πολύ σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορου τομεί. Είχα όμω ε, κάποιε ερωτήσει και αμφιβολίε όταν είχατε πει ότι θα ολοκληρωθούν όλα στις 26 Νοεμβρίου. Σω τα καταφέρετε, είμαι αισιόδοξη. Αλλά βλέποντα του όρου υπό τους οποίους εξετάζουμε αυτά τα θέματα και το DNA και την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί ή να υπάρχει ένα ιδιαίτερα στενό πλαίσιο. Μπορεί ίσω να εξευρεθεί ένα καλύτερο, μια καλύτερη οδό προ τα εμπρό. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε πώ θα λειτουργήσει το χρονοδιάγραμμά σα όλων τούτων λεχθέντων. Αυτέ οι ερωτήσει από πλευρά μα. νομίζω οι συνάδελφοι σε σχέση με αυτό θα το έβρισκαν θετικό Νομίζω ότι επικοδομητικό θα ήταν, αν δεν μπορέσετε να απαντήσετε φυσικά σε όλες αυτές τις απαντήσεις, να μπορέσετε να απαντήσετε ιστερότερα στο έγγραφο που θα μας διαθέσετε. Φαντεν Καμπ παρακαλώ να απαντήσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα γι' αυτό να πω ότι όπως και ο κύριος Φαντάικ και εγώ είμαι Ολλανδός και εδώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε πάντα σύντομοι και είμαστε γνωστό, γνωστοί γι' αυτό οι Ολλανδοί. Με ενδιαφέρον διαβάσαμε αυτή την πρόταση των δύο βασιλείων προσβλέπουμε και αντιμετωπίζουμε αυτές τις ε, προτάσεις με ιδιαίτερη κατανόηση και συμπάθεια. Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις. Η διαπίστευση πρώτον επιτυγχάνεται, γίνεται μέσω των εθνικών αρχών διαπίστευσης. Έτσι, λάβατε υπόψη επίσης και μια ευρωπαϊκή διαπίστευση. Πρώτη ερώτηση, μια και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, όπου χρειάζεται οπωσδήποτε μια ισορροπία μεταξύ προστασίας ε, της ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών προσωπικών ιδιωτικών δεδομένων. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι και εδώ και η πτυχή αυτή τη ευρωπαϊκή διαπίστευση θα διαδραμάτιζε ένα ρόλο. Δεύτερη ερώτηση. Η συνάδελφο ήδη το προανέφερε. Ποιε χρηματοοικονομικέ προσπάθειε θα αναλάβει και θα καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Φαντερκάμ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στις 6.30 όπως προβλεπόταν το έργο μας, τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Και θα έλεγα ότι μπορώ να δω ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που να ζητούν τον λόγο τώρα. Ίσως έχουμε κάποιο λεπτό ακόμα αν θέλει η Σουηδική Προεδρία να κάνει κάποια τελική παρατήρηση. Θα πρότεινα όμως, μια και πολλές ερωτήσεις ε, διατυπώθηκαν και τέθησαν επί και θίγησαν, ίσως θα υπάρχει κάποια ευκαιρία η Σουηδική Προεδρία να απαντήσει γραπτά αυτές τις ερωτήσεις υστερότερα στο εγγύς μέλλον. Μια και δεν υπάρχει κάποια προθεσμία που να έχει τεθεί από το Συμβούλιο ώστε η Ευρωβουλή να ε, ολοκληρώσει τη γνωμοδότησή της. Ίσως αν μπορούσατε λοιπόν να κάνετε κάποια καταληκτική παρατήρηση με χαρά θα την ακούω. 20 Νοεμβρίου είπατε καταληκτική, 26, 26 Νοεμβρίου. Θα υπάρχει λοιπόν καταληκτική προεδρία, υπάρχει, ε, προθεσμία με συγχωρείτε, υπάρχει. Θέλετε να πείτε κάτι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που υποβάλλατε, αναφέρομαι σε όλους τους συναδέλφους. Θα είμαι πολύ σύντομη, θα προσπαθήσω όντως να σας δώσω μια γραπτή λεπτομεριακή απάντηση. Το πιο σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με το ότι η διαπίστευση αυτή καθ' αυτή γίνεται από φορείς διαπίστευσης. Και σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διαπίστευση, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διορίσει μια εθνική αρχή η οποία θα λαμβάνει τι αρμοδιότητε από το κράτο και θα είναι υπεύθυνη για τι διαδικασίε διαπίστευση. Και στη συνέχεια οι αρχέ αυτέ, οι φορεί αυτή διαπίστευση, θα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Διαπίστευση, η οποία με τη σειρά τη είναι υπεύθυνη για να εξασφαλίσει ότι η διαπίστευση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώς έχει όμως η κατάσταση σήμερα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο και που δίνουν μια γενική εικόνα των πραγμάτων δείχνουν ότι όσον αφορά το DNA υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολλούς και διάφορους πολλά και διάφορα εγκληματολογικά εργαστήρια και έχουν ουσιαστικά δώσει διαπίστευση σε αρκετά στα πιο σημαντικά τέτοια εγκληματολογικά εργαστήρια. Όσον αφορά όμως τα δαχτυλικά αποτυπώματα, η διαδικασίες αυτές πολλές φορές έχουν περάσει στις αστυνομικές αρχές, σε άλλους χορούς, σε άλλους φορείς με και διαπίστευση υφίσταται για ορισμένα εργαστήρια αλλά όχι σε όλα σίγουρα. Όσον αφορά τώρα τη συγχρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα να υποβληθούν αιτήσει χρηματοδότησης σχεδίων τα οποία θα έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις ικανότητες του προσωπικού των εργαστηρίων αυτών κτλ. Το βασικό χρηματοδοτικό όμως βάρος θα φέρουν τελικά τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή αυτής της απόφασης. Ο πρόεδρος του ΕΝΦΑΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, συμμετείχε στο σεμινάριο που έγινε στη Στοκχόλμη τον Ιούνιο Καθώ επίση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευση, και συνεχίσουμε εμείς να δίνουμε πληροφορίε προς τους φορείς αυτούς. Η ομάδα εργασία συνεδρίασε όντω τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο και θα συνεδριάσει και αύριο προκειμένου να συζητήσει περαιτέρω αυτό το ζήτημα. Ίσως να αρκούν αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σαφώς και αρκούνε και θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, όπως είπατε, στη γραπτή σας απάντηση. Η Αντιπρόεδρος, κυρία Ίντιβελτ, όμως θέλει τώρα το λόγο. Like... Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως να μην κατάλαβα καλά, αλλά πόσο ξέρω δεν είχε μπει ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίσημη διαδικασία διαβούλευσης και περιμένετε από εμά σε δύο μήνες να υποβάλουμε επίσημα τη γνωμοδότησή μας. Ποιο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να απευθυνθώ βέβαια στη γραμματεία του Συμβουλίου. Έχω ενημερωθεί ότι η Κορεπέρ ζήτησε γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Ιουλίου και ότι η πρόταση δημοσιεύτηκε στην επίση εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να υποβάλει την νομοδότησή του 26 Νοεμβρίου. Θα έρθω όμω πάλι σε επαφή με τι αρμόδιε αρχέ Συμβουλίου για να επιβεβαιώσω την πληροφορία αυτή. Αυτή η πληροφορία πάντω δόθηκε στην Προεδρία. Πρόεδρο, θα προσπαθήσουμε και εμεί να ελέγξουμε την όλη διαδικασία, να επαληθεύσουμε ότι όντω ε, ότι, ότι, έτσι έχουν τα πράγματα. κυρία Φώστερ θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, γίνεται μία πρόταση στα μέση Ιουλίου ενώ προκύπτει νέο κοινοβούλιο, νέα θητεία και έχουμε νέου βουλευτέ οι οποίοι πρωτοφτάνουν στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο. Δεν έχουμε καν συνεδριάσει. Περιμένουμε το Σεπτέμβριο και ξαφνικά μα λέτε ότι πρέπει να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα η προθεσμία αυτή είναι πάρα πολύ στενή πάρα πολύ περιοριστική. Είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα και σίγουρα η προθεσμία αυτή δεν είναι καθόλου ρεαλιστική. Και τέλος να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που δώσατε, αλλά χρειαζόμαστε πιο πλήρες πληροφορίες στα ερωτήματά μας. Θα θέλουμε να γνωρίσουμε ακριβώς ποια είναι τα πορίσματα όλων των συνδράσεων που έχουν γίνει στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Again, I, I fully agree with the point... Κύριε συμφωνώ με τα όσα είπε η και αν σας κατάλαβα καλά, ακόμα επεξεργάζεστε το όλο ζήτημα σε ποια ακριβώ διαπραγμάτευση συμμετείχαμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντω όχι στην τελική σα απόφαση. Αν πράγματι το Συμβούλιο εκτιμά την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να μα διαθέτει και περισσότερο χρόνο, προκειμένου να μπορούμε και εμεί εμπεριστατωμένα να γνωμοδοτούμε. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ όλου για τον επικοδομητικό αυτό διάλογο. Θα σα δω πάλι αύριο στι 10 το πρωί. Σα ευχαριστώ για τη συνεργασία σα.